Αρχίζουμε. Buon pomeriggio Καλό σα απόγευμα. Ξεκινάει η συνεδρία τη Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα, μία μικροαλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Ο εισηγητής για τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται για τα γεωργικά προϊόντα, η Ράτσε Γκαρσία Περές, και ο συνάδελφος Κάπουλα Σάντος, του οποίου το θέμα θα συζητηθεί αύριο, πρέπει να φύγουν νωρίτερα. Οπότε, προτείνω να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη και να ξεκινήσουμε αύριο το πρωί με τα σημεία 11 και 12 και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά. Ανακοινώσεις του Προέδρου αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο η σημερινή μας συνεδρίαση. Όπως ε, ξέρετε συνάδελφοι, τα σχέδια έκθεσης για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, οι αντιπροτάσεις, αυτό που μας αρέσει να το ονομάζουμε έτσι, θα παρουσιαστούν στις 18-19 Ιουνίου. Θέλω λοιπόν να αναγγείλω ότι η προθεσμία για την ε, παρουσίαση τροπολογιών όπως συμφωνήθηκε και με τους συντονιστές είναι 9 Ιουλίου στις 12 για τις άμεσες πληρωμές και τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ ενώ για την, ε, ενιαία, για την ενιαία οργάνωση αγοράς για την ΗΠΕΘΡΟ έχει προβλεφτεί στις 10 Ιουλίου στις 12. Αυτές είναι οι προθεσμίες για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν επί των προτάσεων της Κομισιόν και όχι επί των προτάσεων των εισηγητών. Καταλάβατε. Ξεκινάμε με το σημείο 3. Παρουσίαση της μελέτης πώς να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την αηφόρο καινοτομία στο γεωργικό τομέα. ορίζω τους εμπειρογνώμονες, ε, την καθηγήτρια Janet Dwyer, ε, συνδιευθύντρια του CCRI από το τον Shire. Μετά χαιρετίζω και τον καθηγητή Άλαν Μπάκουελ. Η καθηγήτρια θα παρουσιάσει την μελέτη και ο καθηγητής Άλαν Μπάκουελ θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Ξεκινάει η παρουσίαση. Παρακαλώ. Κύριε Ντουάιερ, χαιρετίζω και τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Πλέμπα, για την παρουσία σου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας και ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε στο Κοινοβούλιο. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και για μένα είναι πολύ εντυπωσιακό. Χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα το απόγευμα και να αναφερθώ στη μελέτη που κάναμε. Θα μιλήσω περίπου για 20 λεπτά και ελπίζω ότι μετά θα ακολουθήσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σε γενικές γραμμές θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας μιλήσω για το περιεχόμενο της μελέτης και τους στόχους της. Επίσης, εν συντομία, θα εκφράσουμε την προσέγγιση μας και τον τρόπο με τον οποίο ε, εργάστηκαν οι εμπειρογνώμονες ε, μαζί με μένα. Τέλος θα αναφερθούμε στα ευρήματα τα οποία σχετίζονται με τα ήδη γνωστά και σχετικά με την ΚΑΠ και θα κάνουμε και μία αξιολόγηση σε αυτό το πλαίσιο της αναθεώρησης, της προτινόμενης αναθεώρησης της ΚΑΠ και θα κάνουμε και κάποιες ε, συστάσεις. Ε, υπογραμμίζω ότι είναι ακόμα ε, προσχέδια προτάσεων γιατί ακόμα δεν έχει λάβει χώρα αυτή η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε την ε, συμβολή σας έτσι ώστε να ε, δούμε προς τα που θα πρέπει να οδηγηθούμε τελικά όσον αφορά τις συστάσεις. Το περιεχόμενο λοιπόν της μελέτης. Θα αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο της ε, μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης, ο όρος βιώσιμη ανταγωνιστικότητα είναι ένας όρος ο οποίος θεωρείται σημαντικός στόχος της πολιτικής. Είναι ενδιαφέρον ε, ότι σε αυτήν την ανακοίνωση το περιεχόμενο ή αν θέλετε τα συμφραζόμενα ε, του ε, όρου αυτού είναι περισσότερο η γεωργική οι γεωργικοί το, η δεύτερη αναφορά μου είναι κάτι που είπε ο Επίτροπος κ. Σιόλος, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιανουάριο του 2011 εκεί συνέδεσε ε, την, ε, ε, την πρόκληση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ σε σχέση και σε διασύνδεση με τις κλιματικές και άλλες περί προκλήσεις και επίσης αναφέρθηκε και στην ανάγκη να διατηρηθεί η χωριακή ισορροπία. Ε, αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο μια δέσμευση έτσι ώστε <clears throat> να γίνει σωστή και ενεργητική διαχείριση ε, της ε, χωροταξίας. Εμείς θελήσαμε να πάρουμε τους στόχους που έθεσε σαν τέτοιους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε κατά πόσον με τα προτινόμενα μέτρα μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα εργαλεία τα οποία έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, λαμβάνοντας επίσης, επίσης και την επιχειρηματολογία των αλλαγών, τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και βλέποντας όχι μονάχα την ΚΑΠ αυτή καθεαυτή, αλλά ε, και τις άλλες διασυνδεόμενες ε, πολιτικές ε, που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτήν την βιώσιμη ανταγωνιστικότητα γιατί βεβαίως ο στόχος ε, είναι να στηριχτεί κατά κάποιο τρόπο η θέση που θα εκφράσει εν τέλει η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο μελετήσαμε έγγραφα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Προσπαθήσαμε να πάρουμε παραδειγματικά χώρες οι οποίες εκπροσωπούν και το Βορρά και το Νότο, μεγάλες χώρες, μικρότερες χώρες, μεγάλες χώρες οι οποίες είναι καθαροί συμβολή στο προπολογισμό κτλ. Επίσης κάναμε και ειδικέ μελέτες περιπτώσεων βάσει στοιχείων ε, των νέων προτάσεων που ε, μπορούν να εστιαστούν ακόμα καλύτερα στην νέα δέσμη ε, προτείνων. Ας πούμε το μέτρο της διαχείρισης κινδύνων, risk management, το οποίο εισήχθη τώρα. Επίσης εστιάσαμε στην προστιθέμενη αξία, η οποία φαίνεται να είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο της ε, νέας πρότασης. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε με τρόπο ώστε να έχουμε όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως ε, και τον τρόπο χρηματοδότησης ή ε, πολλαπλής χρηματοδότησης που θα υπάρξει για αυτή τη μεταρρύθμιση. Από το Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο διήρκεσε η μελέτη Είχαμε πολλούς εμπειρογνώμονες ε, από όλα τα κράτη-μέλη περίπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως θα αναγνωρίσετε κάποια από τα ονόματα. Θέλαμε να έχουμε ε, πραγματογνωμοσύνη και από τα παλιά και από τα νέα ε, κράτη-μέλη. Ξεκινώντας, να είμαστε σαφείς ε, σχετικά με τους ορισμούς που χρησιμοποίησε στις προτάσεις της ε, η Κομισιόν. Και σε αυτό το ειδικό περιβάλλον, έτσι όπως χρησιμοποιείται από την Κομισιόν, νομίζω ότι ο όρος βιώσιμος ε, σημαίνει περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος, διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα να εξακολουθήσουν να είναι θετικά η ανταγωνιστικότητα δεν χρησιμοποιείται επίσης κατά την άποψή μας με καθαρά οικονομικούς όρους, αλλά προσπαθεί να διασυνδέσει την διατήρηση της βιωσιμότητας της γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν αναφέρεται μονάχα στην προώθηση των πιο ε, ανταγωνιστικών ή πιο κερδοφόρων, ας πούμε, εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ε, πρόταση υπάρχει μεγάλη διασύνδεση με την καινοτομία στην Ευρώπη ε, που αποτελεί έναν ε, στρατηγικό, ένα κεντρικό μηχανισμό και για την επίτευξη των νέων στόχων στην γεωργία που θα είναι πιο ανθεκτική, πιο βιώσιμη, που θα είναι σε θέση καλύτερα και αποτελεσματικότερα να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Επομένως, οι οικονομικοί στόχοι, οι κοινωνικοί στόχοι και ε, ε, περιβαλλοντικοί στόχοι διασυνδέονται εδώ. Βλέποντας την μέχρι τούδε εμπειρία, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, στοιχεία τα οποία μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Διαπιστώνουμε πάντως ότι στον ε, τομέα των άμεσων ε, πληρωμών και των μέτρων ε, αγοράς, εκεί έχουμε πιο γενική αντιμετώπιση. Αυτός είναι ο πυλώνας 1 που στηρίζει την γεωργία αλλά χωρίς ιδιαίτερα στοχευμένο τρόπο. Συγκριτικά, οι μηχανισμοί του πυλώνα 2 των υφιστάμενων μηχανισμών έχουν στόχο περισσότερο την προώθηση αυτών των στόχων, ε, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα ε, και επίσης να αντιμετωπίσουν και κάποια ειδικά προβλήματα και επομένως να αντιμετωπίσουν και την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας και ε, ενδεχομένως από εκεί να προκύψουν νέα οικονομικά αλλά και κοινωνικά ε, ε, συγγνώμη, οικονομικές και κοινωνικές βελτιώσεις. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει και μία διαφορά ανάμεσα από τις προσδοκίες του πυλώνα 2 και όσων μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί. Ξέρετε, όταν είναι πολλαπλή η στόχη, βλέπουμε καμιά φορά ότι υπάρχουν ας πούμε δύο προγράμματα τα οποία στην ουσία ενώ βρίσκονται στον ίδιο πυλώνα μπορεί να δουλεύουν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό το διαπιστώσαμε σε αρκετές χώρες. Το πρόβλημα με την μη στοχευμένη βοήθεια ε, είναι ότι δεν καταφέρνεις τελικά να επιτύχεις μεγάλη προσθετικότητα. Τα προβλήματα με τον ε, πυλώνα 2 βεβαίως οφείλονται και, στην και στο ε, γενικότερο σχεδιασμό. Πολύ ε, σοβαρά θα πρέπει να σκεφτούν οι υπεύθυνοι για τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα, τι θέλουμε να επιτύχουμε μέσω της δαπάνης των χρημάτων ή της χρήσης των χρημάτων αυτών. Πρέπει να είναι πιο στοχευμένες οι προσδοκίες. Θα δώσω κάποια παραδείγματα, ας πούμε, ε, projects ε, τα οποία, από τα οποία μπορούμε να μάθουμε. Οι διαδικασίες ε, είναι καινοτόμες και μπορούν να προωθήσουν στοχευμένη έτσι, βελτίωση στον πυλώνα 2. Ας πούμε, ε, βελτίωση της κατανόησης περιβαλλοντικών προβλημάτων, διαχείριση των ε, ε, πόρων της υπαίθρου μέσα στα πλαίσια της πολυλειτουργικότητας, οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Πολλαπλά προτερήματα από κάτω προς τα πάνω, μέσω οργανικής γεωργίας, μέσω ε, βοήθειας που παρέχεται στους εμπλεκόμενους φορείς που ενδεχομένως έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Δεν θα πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Σε σχέση λοιπόν με την επίτευξη της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, καταλήξαμε ότι υπάρχουν πολλά ε, πολλά στοιχεία στην, ε, στις στα προτινόμενα μέτρα που τελικά αποκινητροδοτούν ας πούμε τους ενδιαφερόμενους και επομένως δεν μπορούν τελικά να επιτευχθούν πολλά με τα ε, ενωσιακά χρήματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι και ο ιδιωτικός τομέας επενδύει στην γεωργία και βλέπουμε πολύ προσεκτικά τι γίνεται και ξέρουμε ότι Γενικώ δεν θέλει ο ιδιωτικό τομέα να κάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Θέλει ε, ε, βράχοι πρόθεσμες με άμεση ε, απόδοση ή τέλος πάντων δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις οι οποίες θα προκύψουν στο μέλλον όσον αφορά τις νέες καλλιέργειες, όσον αφορά την τροποποίηση της αντιμετώπισης της υπαίθρου. Βλέπουμε λοιπόν όλα τα προγράμματα αυτά και τελικά ε, βλέπουμε ότι στην ουσία δεν κάνουν παραπάνω πράγματα από αυτό που κάνουν οι τράπεζες όταν χρηματοδοτούν τον γεωργικό τομέα γιατί δεν θέλουν να πάρουν κανένα ρίσκο. Επομένως πρέπει οπωσδήποτε ε, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επενδύσουμε, συγγνώμη, ε, να δώσουμε κίνητρα σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε την πρόοδο σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, πιστεύω ότι ο καθένας δουλεύει ακόμα μόνος του σε έναν εξειδικευμένο τομέα. Ένας δουλεύει για την ε, περιβαλλοντική ε, βιωσιμότητα, ένας άλλος για κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει η ε, σωστή ανάδραση που πρέπει να υπάρχει. βλέποντας επίσης και άλλα στοιχεία ε, στρατηγικής και πολιτικής ε, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν ε, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Βλέπουμε ότι μπορεί να επηρεαστεί ας πούμε η γεωργία και από την έρευνα και την ανάπτυξη και από την πολιτική καινοτομία γενικότερα και επομένως θα πρέπει το πεδίο εφαρμογής, η εμβέλεια να αυξηθεί. Επίσης, κατά την άποψή μας ε, ε, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο πυλώνας 2 έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι πολύ περισσότερο από ότι ε, αν χρησιμοποιηθεί ο πυλώνας 1. αλλά συχνά εξακολουθεί να γίνεται λόγος για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν ας πούμε, αυτά τα ενδεχόμενα. Δύο λόγια θα πω ακόμα γι' αυτό. Βλέποντας τις νέες προτάσεις, ε, μπορώ να σας πω ποια είναι τα συμπεράσματα μου σε αφορά την αξιολόγηση των προτάσεων. Ε, ο, ε, ο, ο, ο πυλώνας 1 αναφέρεται στη στήριξη του εισοδήματος. Δεν είναι όμως μεταποιητικός κατά κάποιο τρόπο μηχανισμός από την ίδια του τη φύση. Η αίσθησή μας λοιπόν είναι ότι βεβαίως μπορεί να παίξει ρόλο ε, στο να ε, ε, επιτευχθεί η χωρική ισορροπία αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα. Στον πρώτο πυλώνα επίσης έχουμε αναφέρει για κάποια άλλα στοιχεία, ε, ας πούμε το Farm Advisory Service ε, και την ε, δυνατότητα της διασταυρούμενης ερεσιμότητας. Εκεί μπορούμε να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και οι επιλογές ε, ε, πρασινίσματος ε, της οικονομίας είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω. Πάντα σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Επανέρχομαι στον πυλώνα 2 λέγοντας ότι το δυναμικό του πυλώνα 2 είναι μεγάλο, είναι μεγαλύτερο σίγουρα από τον πυλώνα 1, έχει ε, πολλές θετικές ε, εξελίξεις και μπορεί καλύτερα να ανταποκριθεί στο μέλλον στο στόχο της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας. Ε, έχουμε εδώ το EIP, το οποίο είναι σημαντικό. Επίσης, ε, μια ευρύτερη ε, συνεργασία και βοήθειες οι οποίες βασίζονται σε ευρύτερη συνεργασία και όχι σε στεγανά ας πούμε, και καθορισμένα στοιχεία. Βεβαίως, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί ο ένας ή ο άλλος πυλώνας μονάχα. Δεν μπορεί δηλαδή με μεμονωμένες κινήσεις να επιτύχουμε την πραγματική βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει η διάσταση, το χάσμα, ανάμεσα στις προτάσεις και την ε, υλοποίηση, τις προτάσεις και την ε, τελική επίτευξη των στόχων δηλαδή. Υπάρχει μια νέα λογική σε αυτές τις προτάσεις, σε σύγκριση με την τροχιά των μεταρρυθμίσεων που ακολουθήσαμε στο παρελθόν. Από τις μεταρρυθμίσεις Μαξάρη 1992 μέχρι τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις και την ενδιάμεση αναθεώρηση Health Check βρισκόμαστε στην τροχιά αποσύνδεσης ε, της υποστήριξης και αναθεώρησης. Άλλαξε η μερίσια διάταξη με αυτό το πακέτο μέτρων, διότι η κυριότερη ιδέα σε αυτό το πακέτο μέτρων είναι η ισοδίκαια κατανομή και η δικαιοσύνη όσον αφορά τα μέτρα από τα κράτη-μέλη και την κατανομή των πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό έχει γίνει η πριτανεύουσα σκέψη ως θέμα στο νέο πακέτο μέτρων. Μπορεί να συζητήσει κανείς και να πει αν χρειάζεται αυτό υπάρχουν σαφή κριτήρια για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή. Και σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν σε κάθε πυλώνα Πιστεύω ότι είναι σαφές ότι ενώ στο παλαιό πρότυπο ο πυλώνας 1 ήταν η υποστήριξη ε, εισοδήματος, ενώ ήταν η αντιστάθμιση όσον αφορά το χάσμα εισοδημάτων και το, ο πυλώνας 2 για την ανάπτυξη της υπαίθρου, στο νέο πακέτο βλέπουμε στοιχεία ανάπτυξης της υπαίθρου και στους δύο πυλώνες και στοιχεία υποστήριξης του εισοδήματος και στους δύο πυλώνες. Παράδειγμα, στοχοθέτηση υποστήριξης νέων γεωργών στον πυλών αυτών που αφορά και την αηφορία, την βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και την αηφορονάπτυξη. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι για τον πυλώνα 2 έχουμε μια διασφάλιση, ας το πούμε έτσι, εισοδήματος, μέτρα διασφάλιση συνολικά. Η εντύπωσή μας για αυτή την αρχιτεκτονική δομή είναι ότι είναι ένα συνεκτικό νέο πρότυπο. Ανησυχούμε όμως μήπως δεν είναι επαρκές μήπως είναι ανεπαρκές για να αλλάξει αυτή η, να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαφορά φάσης με τις νέες προτάσεις. Υποβάλλουμε κάποιες συστάσεις λοιπόν και αυτό είναι εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο να σας μιλήσω σήμερα γι' αυτό και να ακούσω τις απόψεις σας. Μία εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι ότι αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε το μέλλον της ΚΑΠ, κοινή αγροτικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση που τίθεται στον πρώτο πυλώνα και τις επιπτώσεις της ανακατανομής ε, κονδυλίων σε σχέση με τα διάφορα ίδια εκμεταλλεύσεων κτλ. Ο πυλώνας 2, η ανάπτυξη πέθρου σχεδόν χάνεται από τον ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας, όμως είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τις μελλοντικές προσαρμογές και την ανθεκτικότητα και γι' αυτό προτείνουμε ίσως, αν τα κράτη-μέλη είχαν μια πιο συνεπή και συνεκτική, ας το πω έτσι, αναγνώριση της αξίας του πυλώνα 2 στο πακέτο μέτρων, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να αυξηθεί η εστίαση στο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σε σχέση με αυτά, απλά Συνέταξα ένα σύντομο σχέδιο κειμένου εχθές. Στις γραπτές μας προτάσεις προτείνουμε να υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι όσον αφορά τις δυνατότητες για τον πυλώνα 2 από τα κράτη-μέλη. Και αυτό θα σας δώσει μια δυνατότητα να δείτε σε σχέση με τις δαπάνες εφ' εξής, ότι όλα τα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτές τους τις δαπάνες από τα βέλη από την αριστερά για, τον, για το κατόφλι λένε τουλάχιστον 30 ή 40%. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε αυτό έχει επιπτώσει στα παλαιά κράτη-μέλη. Στο να ζητείτε από αυτά να αυξήσουν το ποσοστό της συνολικής ε, κατανομής κονδυλίων για την ανάπτυξη του υπαίθρου, ώστε εκείνοι που θα πρέπει περισσότερο να προσαρμοστούν είναι η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία, το Βέλγιο, σε κάποιο βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο, και προφανώς αν ανοίξουμε ακόμα, αν ανεβάσουμε τον πύχη περισσότερο και άλλα κράτη-μέλη. Η εντύπωση που έχω σε σχέση με αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή τα νέα κράτη-μέλη, πολλά από τα νέα κράτη-μέλη, έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου από ό,τι σε άμεσες πληρωμές και κάνουν λόγο για το μέλλον παράλληλα με κράτη-μέλη για τα οποία τα μέτρα, τα κονδύλια για την ανάπτυξη υπαίθρου είναι ένα μικρό ποσοστό του συνολικού πακέτου. Γι' αυτό είναι δύσκολο να διεξαχθεί μια συζήτηση συγκριτικά για τον ρόλο αυτών των δύο πυλώνων εφ' Αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι η πρώτη μου πρόταση. Ενδιαφέρομαι για τι αντιδράσει σα. Το δεύτερο είναι η μάθηση, η συναγωγή συμπερασμάτων. Και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτό αυτές τις προτάσεις να μετρήσουμε το αποτέλεσμα σε σχέση με τους στόχους, να συναγάγουμε τα συμπεράσματα και να μάθουμε τα συμπεράσματα από αυτή την εποπτεία για αυτές τις επιδόσεις σε μια μεσοδιαστηματική, ενδιάμεση αναθεώρηση σε σχέση με τα μέτρα αυτού του πακέτου. Είναι σημαντικό να υποπτεύσουμε και να επιτηρήσουμε να δούμε ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα ως επιδόσεις. Από, την, ε, από τη μελέτη των επιπτώσεων στα κράτη-μέλη θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερες ρήτες ασφάλειες, ασφάλειας για την α, βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Δεν θέλουμε να πούμε με αυτό ότι υπονομεύεται το περιβάλλον με τα κονδύλια και τα μέτρα που λαμβάνονται τώρα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι για το σχεδιασμό επενδύσεων πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μακροπρόθεσμα την αηφορία. Να μην εντάξουμε κονδύλια σε κάποια πράγματα που μετά από πέντε χρόνια δεν θα έχει νόημα να συνεχιστούν και δεν θα έχουν αποτελέσματα, διότι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά π.χ. τι κλιματικέ αλλαγέ δεν θα αντιμετωπίζονται. Βρήκαμε επίση και κάποια πολύ καλά παραδείγματα όπου οι εμπλεκόμενοι έπρεπε να μπορέσουν να αναπτύξουν τα κριτήρια της στοχοθετημένης συνδρομής ώστε να παίρνουν οι περισσότερο ανα, αναγκαιούχοι, οι περισσότερο αναγκεμένοι αποδέκτες αυτά τα κονδύλια. Σε σχέση και με τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν με τη μέθοδο του όποιος ήρθε πρώτος παίρνει κονδύλια είναι πολύ δύσκολο στο τέλος τέλος έτσι να ταυτοποιήσουμε τι γίνεται. Διότι δεν υπάρχει στοχοθέτηση για τις επενδύσεις για τους περισσότερο αναγκεμένους. Για εκεί όπου θα υπήρχε η ανάγκη υποστήριξη για τους περισσότερο αναγκεμένους. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να πούν εντάξει αυτά τα κονδύλια έχουμε όποιος ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση να υποφεληθεί. Πρέπει να το δούμε λοιπόν διαφοροποιημένα σε σχέση με τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Αν υπάρχει ένα καλό θετικό σχέδιο, ένα πρόγραμμα σχεδιασμού που να μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα θετικά για την επίτευξη των στόχων της Επιτροπής. Συνιστούμε επίσης μια διευρυμένη, έναν διευρυμένο συντονισμό με τα άλλα στοιχεία πολιτικών που είναι και αυτά σημαντικά και υπησερχόμεθα σε αυτά ως στοιχεία σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην έκθεσή μας για τις συστάσεις τώρα σε σχέση με τον πυλώνα 1 για τις προτάσεις για άμεσες ε, πληρωμές περισσότερο από ό,τι για διαχείριση των αγορών όπως προανέφερα θα θέλαμε να είναι πιο ενδυναμωμένος ο ρόλος όσον αφορά τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Αυτό θα έχει κέρια σημασία όχι μόνο για τα νέα κράτη-μέλη αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν αρκετές μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς πόρους στο μέλλον. Ιδιαίτερα όταν σπανίζει το νερό, οι ε, υδάτινοι πόροι, όταν έχουμε μόλυνση ε, εδαφών κτλ. Να κατανοήσουμε αυτές τις επιπτώσεις και πραγματικά να σχεδιάσουμε επιτυχείς στρατηγικές για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα στο μέλλον θα έχει κέρια σημασία ως δράση. Και θεωρούμε ότι το εύρος ε, πρέπει να διευρυνθεί η εμβέλεια, να επεκταθεί περισσότερο για την αξιολόγηση που έγινε πριν από λίγα χρόνια βρήκαμε ότι μειονότητα μόνο των γεωργών επιτυγχάναμε ως στόχους ε, και δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί ευρύτερα. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα στενά πλαίσια και να επεκτείνουμε το φάσμα. Όσον αφορά τις προτάσεις πρασινίσματος, greening, είναι δύσκολο να πει κανεί ε, ποια συμφωνία θα επιτεθεί τελικά, αλλά θα υπάρξει κάποιο περιθώριο τα κράτη-μέλη να ασκήσουν τη διακριτική του ευχέρεια σε κάθε, κάποιο βαθμό για την χρήση των κονδυλίων. Αν συμβεί αυτό, θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να επεξηγήσουν τι επιλογέ που θα κάνουν ή που θα έχουν κάνει όσον αφορά το πρασίνισμα του πυλώνα πληρωμών. Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα μπορούμε να μάθουμε μαθήματα, να συνεργάσουμε συμπεράσματα από αυτό. Και μετά ερωτήματα ποια θα είναι τα κριτήρια στο μέλλον για τον πυλώνα 1. Πώς θα πρέπει να κατανέμεται η συνδρομή μεταξύ κρατών μελών. Και αν συμβαίνει ότι η στόχη να έχουμε περισσότερους πυλώνες θα οδηγήσει σε μια συνεκτικότητα δομών και διαρθρώσεων, δεν θα πρέπει να υπάρχουν πιο συνεκτικά κριτήρια συγκρίσιμα μεταξύ τους για την κατανομή αυτών των κονδυλίων. Κάποιες εξειδικευμένες συστάσεις για τον πυλώνα 2. Χρειαζόμαστε κάτι πιστεύω, για να μας δώσει την δυνατότητα η διοίκηση, οι υπάλληλοι, οι φορείς για τις πληρωμές στα κράτη-μέλη να αισθάνονται ότι πρόκειται για μια μεταμόρφωση πραγματικά, για μια αναδιάρθρωση. Δεν είναι μόνο να διαθέτουμε κονδύλια για εκείνους που θα κάνουν επενδύσεις ούτως ή άλλως. Είναι να προσπαθήσουμε μακροπρόθεσμα να δούμε τα πράγματα, να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που θα γινόταν με τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να τα σκεφτούμε σε βάθος προσεκτικά. Οι συστάσεις μας είναι ότι η βοήθεια, η συνδρομή θα είχε μεγαλύτερα αποτελέσματα αν μέσω μιας τοπικής στρατηγικής θα μπορούσε να κατανέμεται για τις αποφάσεις τι είναι σημαντικό. Ίσως μια υποκατηγορία για την ε, γεωργία ή για τις ε, επιμέρους διαθρώσεις, δια, ε, διασύνδεση μεταξύ προϊόντων, διάθεσής τους, πρωτο, τουριστικών πρωτοβουλειών και μιας ημερήσιας διάταξης ατζέντα για την ανάπτυξη ανάπτυξη των περιφερειών, των χώρων της υπαίθρου. Είναι περίπλοκο να τα κάνει κανείς αυτό, αυτά και να τα σχεδιάσει. Και αυτό ίσως αφ' αυτού θα μπορούσε να ήταν ένα αρνητικό κίνητρο. Είπαμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα, να μπορούν να εμπλέξουν μεγαλύτερα κονδύλια, να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και για τη χρήση αυτών των κονδυλίων, θα συνεισέφερε να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκαμπτες ή ε, αυτές τις δυσκολίες ή ακαμψίες. Θα θέλαμε να δούμε ότι θα πετυχαίναμε μεγαλύτερη, ας το πω έτσι, ε, κατευθυντικότητα ε, συνάγοντας ε, παράλληλες ε, δράσεις με το leader όπου εδώ οι κατευθυντήριε γραμμέ και οι προσανατολισμοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σημαντικό στοιχείο για το leader σε σχέση με το τοπικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε κάτι τέτοιο. Ίσως όχι την ίδια ταυτόσημη δομή, αλλά κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα εφάνταστα να δράσουν, να εμπνεύσουμε του πολίτε, να έχουμε κάτι καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα, με πιο εφάνταστε δράσει. Θετικό θα ήταν αυτό. Εδώ βλέποντα πάλι τα προσκόμματα για την καινοτομία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σχέση με τον ευθυγραμμισμό ή σύγκληση των κανονισμών και ρητρών για τα διαθωτικά ταμεία, αν δούμε την στρατηγική μας στοχοθέτηση για τα κονδύλια σε τοπικό επίπεδο, είναι αξιοπερίεργο μας φαίνεται ότι ο κανονισμός για την ανάπτυξη της υπαίθου θα έπρεπε να έχει πιο αυστηρούς κανονισμούς και ρήτρες από ότι σε άλλες δράσεις. Αυτό θα αποτελούσε πρόσκομα όσον αφορά την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν οι πολίτες και έχουμε και την δυνατότητα ε, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επικεντρωνόμαστε σε συμβουλές, σε πληροφορίες, δίνοντας στους πολίτες πραγματικά την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να δοκιμάσουν και να δοκιμαστούν σε αυτές τις δράσεις στο τοπικό επίπεδο. Και πρέπει να δούμε κατά πόσον η χρηματοδότηση αυτή θα μπορούσε να εμπλέκει και την αντιμετώπιση κινδύνων με βάση όλα αυτά. Αυτά είχα να αναφέρω και ολοκληρώνω. Ίσως ότι θα ήταν, ότι είναι επικοδομητική αυτή η παρουσίασή μου και αναμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Προχωράμε στις ερωτήσεις. Εγγράφτηκαν διάφοροι συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την ε, Μπρίτα Έγμενς και μετά με την Έλγα Τόρφμαν. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης. Ήταν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις μεταξύ άλλων. Μεταξύ αυτών βρήκα ενδιαφέρον ότι είπατε ότι με τα δημόσια κονδύλια πολύ σπάνια τολμούμε να ρισκάρουμε κάτι και να υπομισθούμε κάποιους κινδύνους και να είμαστε καινοτόμοι. Τι θα γινόταν αν για παράδειγμα προσπαθούσαμε, μια και πρέπει να είμαστε όλο και πιο αποτελεσματικοί στην χρήση αυτών των κονδυλίων, προσπαθούσαμε τα κονδύλια αυτά περισσότερο στο χώρο της υπαίθρου να τα εμπλέξουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε ανακυκλούμενα με τις ε, πιστώσεις και τα δάνεια αυτά να επιτρέψουμε δράσεις ε, όπου εδώ και αν θα γινόταν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη περιφέρειες για τους φορείς ή κομβικά σημεία ε, κατανομής ώστε να υπάρχουν και κάποια ποσοστά που θα λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία διαφορετικά δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν τόσο εύκολα. Θα πρέπει να αποδεικνύουν την βιωσιμότητά τους οικονομικά αυτά τα ε, προγράμματα. Αλλά ένα ποσοστό ουσιαστικά εγκρίνεται ώστε να ξεκινήσουν κάποια νέα προγράμματα και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ή δεν υπάρχει ιδιαίτερη ας το πω έτσι τόλμη ε, θα μπορούσαν κάποια κονδύλια να επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλούμενα. Τι λέτε γι' αυτό. Το χαιρετίζω ότι λέτε σαφώς ότι ο δεύτερος πυλώνας δεν μπορεί να εργαστεί στοχοθετημένα, θα πρέπει πιο στοχοθετημένα να δρά και να ενισχυθεί και χρηματοοικονομικά. Και με ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι είπατε ότι από πλευρά συμβουλών στη Γεωργία πρέπει να δράσουμε ενισχυμένα, διότι στις συμβουλές ή στην διαρροή, διάχυση, διάχυση πληροφοριών, με συγχωρείτε, πολλά περισσότερα μπορούμε να κερδίσουμε κερδίσουμε και να αποκομίσουμε ως ωφέλη. Ίσως και αντίστροφα πάλι το ίδιο. Χρειαζόμαστε σίγουρα τοπικές στρατηγικές επιτόπου. Δεν βοηθάει ισοπεδωτικά από το κέντρο της Ευρώπης, από τις Βρυξέλλες, πανευρωπαϊκά να κόψουμε κοστούμι για όλους τους γεωργούς ισοπεδωτικά. Έχουμε διαφορές μεταξύ μας και πρέπει να λαμβάνονται αυτές υπόψη σε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Σωστό είναι αυτό που είπατε για την ε, εξίσωση προσωμείωση των άλλων ταμείων και καταλήγουμε εδώ και στο θέμα της συγχρηματοδότησης στον χώρο της υπαίθρου. Θα είχαμε αφενός την δυνατότητα με εναλλακτικέ δυνατότητες συγχρηματοδότησης περιοχές και περιφέρειες που είναι οικονομικά δύναμες και δεν μπορούν να διασφαλίσουν τέτοια συγχρηματοδότηση αυτές οι περιφέρειες να μην εξαιρεθούν και βρεθούν εκτός του πλαισίου αλλά να είναι δυνατόν να διεξαχθούν εκεί διαρθρωτικές επενδύσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τις μειονεξίες της, ε, του χώρου της υπαίθρου και θα μπορούσαμε να, να, να βοηθήσουμε να διασ χυθεί λίγο ο κίνδυνος ή το ρίσκο και να βοηθήσουμε για κάποια προγράμματα τα οποία επιθυμούμε να χρηματοδοτηθούν με την μείωση της συγχρηματοδότησης μπορεί να είμαστε πιο λειτουργικοί και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να στεφθεί με επιτυχία ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Ο Χέρμπερτ και μετά ο Μάρτιν Όσλινγκ. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει ακόμα και αν βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε να συζητήσουμε για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, να θέσουμε το ερώτημα. Τι θα γίνει αν υλοποιηθούν όλα αυτά όπως προτείνονται. Το 2020 τι θα γίνει στο τέλος τέλος. Η γεωργία στην Ευρώπη θα είναι ανταγωνιστική ή όχι. Δηλαδή αυτά τα μέτρα θα συνεισφέρουν πραγματικά η γεωργία να είναι πιο ανταγωνιστική στην Ευρώπη ή όχι. Και έτσι θα συνεισφέρουμε η Γεωργία ισχυρότερα να στέκεται αυτόνομα στα ίδια της τα πόδια ή μετά από 7 χρόνια θα πούνε οι Γεωργοί θα, ότι θα έχουν αποδεκτά εισοδήματα. Μπορούμε κάτι τέτοιο να το ε, διασφαλίσουμε. Νομίζω ότι πολύ λίγο θέτουμε αυτά τα ερωτήματα και με την όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση του πρώτου πυλώνα πραγματικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δεύτερη, τον δεύτερο πυλώνα και τη δεύτερη κατεύθυνση. Να υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα για την βελτίωση αυτής της κατάστασης. Κάνουμε λόγο πολύ για την αηφορία και την ενίσχυση της, και ένταση της αηφορίας. Αν δούμε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή, κάποια ερωτήματα αναφύονται. Ένα ε, ακραίο παράδειγμα προτείνεται ένα μέρος, 5%, 7%, 10%, όποιο και ποσοστό να είναι αυτό, της έκτασης για οικολογικές χρήσεις ε, να ε, βρεθεί εκτός ε, εκμετάλλευσης και να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα, έτσι. Δεν θα είναι η οι η ώστε τις πιο εντατικές καλλιέργειες να τις αποσύρουν. Τις πιο δύσκολες για καλλιέργεια αυτές θα αφαιρέσουν ή και τη στην ορεινή Γεωργία τα προβληματικά αυτά ε, σε έκταση ε, τμήματα θα το κάνουν, θα δεχτούν να γίνει αυτό. Και σε σχέση με την, ε, την περιορισμένη έκταση για την μεγαλύτερη εντατικοποίηση εκεί όπου θα απομένει καλλιεργούμενη έκταση, αυτό θα οδηγήσει ώστε η πιο εντατική γεωργία, αυτή που είναι η πιο εντατική στις καλλιέργειες, αυτοί δεν θα διαφερθούν καθόλου για, όλες αυτές, για όλα αυτά τα μέτρα και θα βρεθούν ξαφνικά εκτός, διότι εδώ με την ανώτατα εντατική γεωργία κερδίζουν αυτοί κάποια ε, το εισόδημά τους. Πρέπει εδώ λοιπόν να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Διαπιστώνω και είμαι απόλυτα της ίδιας γνώμης ότι αυτή η βραδία μετάθεση από τον πρώτο πυλώνα στον δεύτερο πυλώνα που τα είδαμε και τα ζήσαμε με 20 χρόνια τώρα ε, χρονοδιάστημα να, και βλέπουμε ότι υπάρχει και διέρεση έχουν κατά 10% ε, κάποια κράτη 70% και μετά κάνουμε λόγο για την δικαιοσύνη στην κατανομή των κονδυλίων στον πρώτο πυλώνα. Ε, ούτε και αυτό μπορεί να γίνει και να δεχθούμε κάτι τέτοιο ως κατάσταση. Και θα έλεγα πρέπει πραγματικά κάποιες ερωτήσεις να θέσουμε. Όλα αυτά συνεισφέρουν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας θα έλεγα αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλω να διατυπώσω. Στο δεύτερο πυλώνα υπάρχει σαφώς το ερώτημα ή ασκείται η επίκριση ότι έχει λένε μεγάλο κίνδυνο όσον αφορά τον πυλώνα 2 από τη γεωργία σε άλλους τομείς. Πράγματι συμβαίνει αυτό. Και πράγματι πρέπει κάποτε να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Αν αρκετά συχνά το βλέπουμε ότι σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα είναι σημαντικά τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα. Τι μπορούμε να κάνουμε, η διολύστηση κονδυλίων να ανασχετηθεί, να μπορέσουμε να ανασχετήσουμε την ε, διαρροή κονδυλίων από τον δεύτερο πυλώνα ώστε να υπάρξει μια πιο αποδεκτή πολιτική και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν. Μάλιστα. Θα ήθελα να ερωτήσω κάποια πράγματα, να θέσω ερωτήματα με κριτικό πνεύμα. Η αηφορία, η, η ε, βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, πληθωριστικά μιλάμε για αηφορία ή για βιωσιμότητα. Τι θα πρέπει στην ανταγωνιστικότητα να ενισχυθεί. Πρέπει πρώτα αυτό να το καθορίσουμε σε έναν ορισμό. Έχω την εντύπωση τα τελευταία χρόνια έχουμε προγράμματα που υποβάλλονται για την προώθηση του ανταγωνισμού στην Γεωργία και να εξωθηθούν εκτός ανταγωνισμού κάποιες επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρξει όμως πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη του ανταγωνισμού σε σχέση με τη Γεωργία και έναντι του τομέα του εμπορίου. Και όχι μόνο να υποστηρίξουμε στην ίδια τη Γεωργία, αλλά να υπάρξουν και διαθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Μια άλλη έννοια χρειαζόμαστε λοιπόν και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από αυτήν που χρησιμοποιούμε. Για μένα θα μπορούσε να είναι αυξημένη, αναβαθμισμένη ποιότητα και αναβαθμισμένη αξία. Αυτό πρέπει να δούμε και για τη γεωργία. Νομίζω συμφωνούμε ότι με τον πρώτο πυλώνα έχουμε λιγότερο στοχοθετημένα δράσεις. Είναι σαφές αυτό. Θα τα αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν μακροπρόθεσμα. Θα λέμε είναι μια υποστήριξη εισοδήματο ή θα υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση και με τα μέτρα του πρώτου πυλώνα. Νομίζω ότι εδώ μπορεί κανεί να το δει έτσι σε σχέση με τις προτάσεις Επιτροπής και είναι θεμητό αυτό. Συμφωνώ μαζί σας όμως ότι για το δεύτερο πυλώνα συζητάμε πολύ λίγο δημόσια και πραγματικά το μεγαλύτερο, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε μεγάλες ανισότητες και ετεροβαρείς σχέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση και μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να καταφέρουμε στο τέλος τέλος να έχουμε την ίδια προσφορά για τα κράτη-μέλη στον δεύτερο πυλώνα, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να ακολουθήσουν την υποστήριξη και ενίσχυση περιβαλλοντικών μέτρων έτσι όπως θα τους τα προτείνουμε να δράσουν και όχι μόνο το θέμα της συγχρηματοδότησης για πολλά κράτη-μέλη που αποτελεί πρόβλημα όλο και περισσότερο για κάποια κράτη-μέλη σε σχέση και με την πρόταση της Επιτροπής που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη ή δεν εξετάζει επαρκώς αυτή την κατάσταση και μάλλον ίσως ε, και επιδεινώνει και τα πράγματα. Θα είχα μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Διαχείριση κινδύνου στον δεύτερο πυλώνα. Τι γίνεται εδώ. Ανοησία αυτό διαχείριση κινδύνου στον δεύτερο πυλώνα, να εντάξουμε αυτή τη διαχείριση κινδύνου στον δεύτερο πυλώνα. Δεν ανήκει εκεί. Άλλες μεθόδους και προσεγγίσεις πρέπει να βρούμε σε σχέση με τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι μη προβλέψιμα τα προγράμματα, τα προγράμματα και οι δράσεις στον δεύτερο πυλώνα όσον αφορά αυτού του κινδύνου, αυτή την πτυχή. Οι συμβουλές, η συμβουλευτική δραστηριότητα πρέπει να ενισχυθεί αλλά πώς θα μπορέσει να γίνει και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Και εδώ αυτό ε, ταιριάζει σε αυτά τα οποία προανέφερα. Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε, ποια γεωργία θα υποστηρίξουμε και πού θα, διατεθούν, θα διατίθενται τα κονδύλια. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Ένα σημαντικό στοιχείο αναφέρατε ολοκληρώνοντας νομίζω, ότι τα προγράμματα leader είναι πραγματικά υποδειγματικά Πολύ λίγο λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα από αυτά τα προγράμματα. Χαιρετίζω λοιπόν να ληφθεί αυτό υπόψη και δεύτερο. Η διαρθρωτική προώθηση σε σχέση με τους νέους, ε, τις νέες κατευθύνσεις το θεωρείτε αυτό σωστό σε σχέση με τους παλαιούς άξονες που είχαμε ακολουθήσει ή νομίζετε ότι δεν πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ο Αλμπερντές και μετά ο Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Δεν είναι απόλυτα σαφές όμως για μένα ποια είναι η στοχοθέτηση, ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της μελέτης. Διότι η στοχοθέτηση ήταν να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και μάλιστα περισσότερο βιώσιμη ή αηφόρο ανταγωνιστικότητα. Ακούγοντας όμως τα όσα μας είπατε, σίγουρα υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις που ήταν σωστές. Είπατε για παράδειγμα ότι ο δεύτερος πυλώνας ε, <clears throat> είναι ενδεδειγμένος, θετικά ενδεδειγμένος, ώστε να πετύχουμε προτερήματα και όσο αφορά το περιβάλλον. Και μετά το χαιρετήσατε από την άλλη πλευρά ότι τα μέτρα του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα συγχέονται και αναμειγνύονται και αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Και θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό αυτά τα ερωτήματα. Και ένα πράγμα στην όλη ε, σύνοψή σας είδα ότι απουσιάζει για την ανταγωνιστικότητα. Γνωρίζουμε ήδη σήμερα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο άσκησε επικρίσεις επ' αυτού ότι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργούν σε μεγαλύτερη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Και η επιβάρυνση αυτή συσχετίζεται σε σχέση με του γεωργού μα, η γραφειοκρατική επιβάρυνση και με τον ανταγωνισμό. Θα ήθελα μια απάντηση από αυτόν. Είχαμε αποφασίσει μέχρι το 2015 από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου να μειώσουμε το γραφειοκρατικό βάρο κατά 20 ή 25% και αντίθετα αυτέ οι προτάσει θα δημιουργήσουν πρόσθετη επιβάρυνση γραφειοκρατική 20%. Αυτές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποτέ δεν θα τύχαιναν της δικής μου υπεψήφισή, Δεν θα, δεν θα δεχόμουν ποτέ να επομισθούν, να ανεχθούν ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατική επιβάρηση οι γεωργοί, οι γεωργοί μας στην Ευρώπη και σε σχέση με την, ε, τη δική μας δράση, στην δική μας ε, εκμετάλλευση και σε σχέση με τη δουλειά που συνεχίζουμε ο γιος μου, εγώ, ακόμα και στις διακοπές, έπρεπε να συμπληρώνουμε όλα αυτά τα χαρτιά, το χαρτομάνι, επιπρόσθετα σε όλα αυτά τα χαρτιά που συμπληρώναμε, για να είμαστε εντάξει γραφειοκρατικά. Ε, και τι θα γίνει, δεν θέλω και του, ας το πω έτσι, και της πεντηκοστής ε, να, να δουλεύω σε αυτή την υποχρεωτική συμπλήρωση ε, δεδομένων και εγγράφων. Θα ήθελα να ξέρω ποια πιο στοχοθετημένη μεταρρύθμιση γεωργική μπορεί να επιτευχθεί, χωρί, χωρίς ε, γραφειοκρατική επιβάρηση. Βλέπω να απουσιάζει ακόμα αυτό το στοιχείο, δεν μας έχει δοθεί. Θέλω να αναφέρω κάτι άλλο που χρειαζόμαστε απαντήσει. Ο Χέρμπερ το προανέφερε. Είπε, αν ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα, και εγώ είμαι απόλυτα υπέρ του να γίνει αυτό και έχω κάθε συμπάθεια και έχουμε και παραδείγματα στην Ευρώπη, Νότιο Τυρόλο, ε, ε, Βαβαρία, Βάδι Βιρτεμβέργη και αλλού, ότι ο δεύτερος πυλώνα εξαιρετικά μπορεί έτσι να λειτουργήσει. Αν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το δεύτερο πυλώνα πρέπει να αποφύγουμε τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται όλο και πιο ενισχυμένα ή να εκραίουν σε μη γεωργικού τομεί και δραστηριότητε. Θέλω να ακούσω τέτοιε προτάσει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε κατάλογο μέτρων που θα καταρτήσουμε και θα θεσπίσουμε για ποιε χρήσει τα κονδύλια του δεύτερου πυλώνα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται. Δεν θα μπορούν έτσι να αποξενωθούν από τη σωστή του ε, εμπλοκή και σωστή του χρήση. Λοιπόν, έχω ανοιχτό πνεύμα για τέτοιε προτάσει, αλλά πρέπει να δούμε και αυτές τις πτυχέ. και για τον Μάρτιν <clears throat> χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω τα προγράμματα, τα σχέδια leader υπάρχουν και πολύ καλά αλλά όταν στη δική μου περιφέρεια βλέπω τα τελευταία χρόνια ε, τα προγράμματα αυτά leader δεν ήταν η συντριπτική του πλειοψηφία για την αηφορία και την ε, μεγαλύτερη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και έτσι δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Θα πρέπει να επανέλθουν αυτά τα κονδύλια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας στη σωστότερη χρήση. Θα ήθελα απάντηση από αυτόν. Ποιες είναι οι επιπτώσεις αν υπάρχει τέτοια ισχυρή ανάμειξη του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Δεν θα ήταν πιο σκόπιμο ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας όσον αφορά τις δαπάνες να διαχωρίζονται κάθετα με σαφήνεια όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου για αυτό που προαναφέρθηκε, είναι σαφές ότι αυτό ανήκει στον πρώτο πυλώνα. Εκεί πρέπει να ενταχθεί και να δούμε πώς από πλευράς των κρατών μελών θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και να χρηματοδοτείται από τον πρώτο πυλώνα τα μέτρα για το περιβάλλον και λόγω μεγαλύτερης ελαστικότητας πρέπει να εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα. Εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε λύσεις για τα προβλήματα ώστε ευρωπαϊκά να χρησιμοποιούνται περισσότερο συγκρίσιμα και με μεγαλύτερη σύγκληση. Και μια άλλη παρατήρηση επιπρόσθετα για την χρήση μεταξύ κρατών μελών και ως Γερμανός Ευρωβουλευτής είμαι υπέρ του οι χώρες εκείνες που απέχουν από το μέσο όρο θα πρέπει να υποστηριχθούν. Εκείνες που βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο θα πρέπει να μην παίρνουν αυτά τα κονδύλια πλέον γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε δίκαιοι για την κατανομή των κονδυλίων στην Ευρώπη και δεν θα είναι υπεύθυνο πια οι ε, γεωργοί να παίρνουν στη βάδια ας πούμε χίποσο και σε σχέση με άλλους ε, που ε, θα έπρεπε να παίρνουν για παράδειγμα ε, περισσότερα. Θα πρέπει εδώ οι αδικίες που υπάρχουν να αντισταθμιστούν και να προσαρμοστούμε στην εκμετάλλευση, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπό οικονομικότερο πνεύμα. Και έτσι θα πρέπει να βρούμε, να εξεύρουμε καλύτερες απαντήσεις για αυτά τα προβλήματα από αυτές που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμως το οποίο ακόμα περισσότερο με ενδιαφέρει και αν σε αυτή τη μελέτη τώρα αυτό αξιολογείται ή όχι, εσείς το αναφέρατε πιστεύω πιο πριν. Είναι οι μεγάλες διαφορές που έχουμε σε σχέση με τα, με τα κράτη-μέλη. Και ο Χέρμπερτ που είναι δίπλα μου και που στο νότιο Τυρόλο παίρνουν από τον πρώτο πυλώνα 50 ευρώ, αλλού παίρνουν 500 ή 600 ευρώ. Αν παραμένει έτσι, παραμείνει έτσι, τότε θα πρέπει να δούμε και την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να υπάρξει μια αντιστάθμιση. αντιστάθμιση. Αυτές οι ε, ανισότητες πρέπει εκεί σε αυτό το πλαίσιο να ε, ρυθμιστούν. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό το θέμα με την ε, ισότητα όσον αφορά τις πληρωμές και την, τις ενισχύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε αυτό. Ευχαριστώ. Grazie, Albert. Ευχαριστώ, Άλμπερτ, ο Τζιμ Νίκολσον και μετά ο Σμιθ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, ομάδα που ήρθε να μας κάνει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και σωστή και ευχάριστη ε, παρουσίαση. Αναφέρθηκαν ε, στο πιο παραγωγικό ε, ε, κομμάτι. Ναι, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν περιοχές που παράγουν περισσότερο και περιοχές που παράγουν λιγότερο. Και όσον αφορά ε, για το γάλα, ξέρετε κάτι για την γαλακτοκομική παραγωγή. Εγώ ήμουν εισηγητής για τον γαλακτικό τομέα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου βεβαίως ε, η κτηνοτροφία ε, στα βουνά είναι σε ορεινές περιοχές είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ λιγότερο παραδοσιακή από την παραγωγή στις παιδιάδες. Ε, το θέμα είναι πώς είναι δυνατόν κάπως να περιοριστούν αυτά τα κενά. Επίσης όσον αφορά τις δυνατότητες ε, του πυλώνα 1 και του πυλώνα 2, ε, αυτό το 30% του πρασινίσματος που προτείνεται στο ε, πυλώνα 1 το είδατε λίγο, είδατε πώς μπορεί να γίνει αυτό και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί στον πυλώνα 2. Είδατε πώς είναι δυνατόν σε αυτή την περίπτωση να επιτύχουμε απλούστευση του συστήματος. Επίσης αναφερθήκατε ε, σε μη στοχευμένες επενδύσεις. Μήπως μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια περισσότερα. Πού ε, σε ποιες περιπτώσεις ε, στα παλιά κράτη-μέλη, στα νέα κράτη-μέλη έχουν γίνει λιγότερο στοχευμένες επενδύσεις ή είπατε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο διευρυμένο πυλώνα 2 σε σχέση με τον πυλώνα 1 Μήπως μπορείτε να αναπτύξετε λίγο τη σκέψη σας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ε, σκέψη αυτή και θα θέλαμε να καταλάβουμε κάπως καλύτερα ε, πώς έχουν τα πράγματα. Και επίσης να δούμε ποια είναι τα επιτυχημένα σημεία από τα οποία μπορούμε να βασιστούμε για το μέλλον. Το μεγάλο ερώτημα είναι όχι πώς θα ανταγωνιστούμε μέσα στην Ευρώπη, αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα ανταγωνιστούμε τον ε, Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου. Αυτό πρέπει να δούμε λίγο και θα πρέπει να το λύσουμε γιατί η αγορά ε, είναι πλέον μεγάλη και επομένως εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε μια αγορά για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Αυτό το Farm Advisory System που λέτε ότι είναι ε, θετικό, πώς το εκλαμβάνετε. Λέτε ότι θα πρέπει δηλαδή να ε, διευρυνθεί, να έχουν περισσότερους συμβούλους, ας πούμε, τα κράτη-μέλη. Από ό,τι καταλαβαίνω, ε, η Κομισιόν λέει ότι ο διαχειριστικός προϋπολογισμός θα είναι αυξημένος και το 15% στα κράτη-μέλη. Επομένως, η ερώτησή μου είναι θυμάμαι ότι στην Ιρλανδία, που είναι η, χώρα μου, η χώρα μου, ε, είχαμε το Farm Advisory Service και τώρα έχουμε το Farm Police Service. Έχουμε δηλαδή ένα αστυνομικό σύστημα το οποίο, που στέλνει τον αστυνομικό από τις Βρυξέλλες. Πώς είναι δυνατόν αυτό να απλουστευθεί. Πώς είναι δυνατόν η δουλειά επιτόπου να γίνει πιο απλή και πιο καλύτερη τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξηγούν επίσης γιατί κάνουν ορισμένε επιλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τζιμ. Ο Σμίχ και μετά ο Άγνιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί καλύφθηκα από άλλους συναδέλφους. Ε, δεν το είχαμε ε, κανονίσει, αλλά νομίζω ότι από, το, την αστυνομική υπηρεσία στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος προηγουμένως ε, θα ξαναπάω εγώ στο advisory service, αυτή τη συμβουλευτική υπηρεσία που μπορεί να βοηθήσει να συμβουλέψει τους γεωργούς για τις επενδύσεις τους, για την αντιμετώπιση που θα έχουν κτλ. Εγώ είμαι παλαιό μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και βεβαίως είναι γεγονός ότι πρέπει να ε, ε, ευθυγραμμιστούν ε, οι κανονισμοί γιατί διαφορετικά υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία τελικά περνάνε μέσα από τις χαραμάδες είτε των αποφάσεων της Κομισιόν είτε των προτάσεων της Επιτροπής μας και κάθε τόσο ζητάμε από τους γεωργούς να κρατάνε τα βιβλία τους με διαφορετικό τρόπο, να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν ε, ρυθμίσει ας πούμε τα πράγματα μέχρι τότε. Έχετε υπολογίσει αυτό το επιπλέον κόστος της συμπληρωματικότητας. Έχετε κάνει κάποιον υπολογισμό. Βεβαίω, στα κοινά στρατηγικά πλαίσια γίνεται μια προσπάθεια να εξευρεθούν ε, λύσεις και βιώσιμες προτάσεις, αλλά παρόλα αυτά ε, εάν έχετε κάνει κάποια αξιολόγηση εσείς που θα μπορούσε να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, θα το εκτιμούσαμε ιδεόντως. Ευχαριστώ πολύ. Άγνιου και μετά σε Κυρίσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μονάχα στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα θα αναφερθώ δύο από τα θέματα της παρουσίαση, δηλαδή. Η καινοτομία δεν είναι κάτι που επιβάλλει στον άλλο. δεν μπορείς να του πεις τώρα θα καινοτομήσεις. Μπορείς απλώς να δημιουργήσεις την ατμόσφαιρα, το υπόβαθρο έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν ε, οι ε, ενδιαφερόμενοι να επιτύχουν καινοτομία. Ε, όσον αφορά δε τον ανταγωνισμό προκύπτει από την βελτίωση και προσαρμογή της ανταγωνιστικότητας. Ε, είδα ας πούμε ε, στην δικιά μου περίπτωση ότι πολλές περιπτώσεις είχαμε βελτίωση της καλλιέργειας των ζαχαροτέφρων και μάλιστα με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Επίσης είδαμε περιπτώσεις όπου μπορεί το έδαφος να έχει, που μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγή και χωρίς ε, αγρανάπαυση και χωρίς ιδιαίτερη αντιμετώπιση του εδάφους. Αυτό δεν είναι καινοτομία. Ε, η ε, λιγότερη χρήση ή η καλύτερη χρήση ή η χρήση διαφορετικών εντομοκτώνων και λοιπόν τέτοιων παρασιτοκτώνων δεν είναι καινοτομία, δεν οδηγεί σε τελικά καλύτερη ποιότητα, καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, θα έπρεπε να είχαν πει ας πούμε ε, και το είπαν εν μέρη σε κάποιες χώρες ότι για να έρθετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνετε μέλη ε, τότε δεν θα πρέπει να κάνετε καινοτομία. Ναι αλλά τι είδους Ευρώπη είναι αυτή επίσης. Πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε επίσης ε, την, ε, ε, τις εμπορικές αρχές οι οποίες μπορεί να επιτρέψουν πούμε, σε κάθε φορτίο γεωργικού προϊόντος να υπάρχουν ε, ο, οτιδήποτε ξένα σώματα μπορείτε να φανταστείτε, χώμα ε, κτλ. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ένας ξένος διαφορετικός σπόρος. Ναι, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν χώρες ή άνθρωποι μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να καταστραφεί η δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα αλλά τελικά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ε, τελικά υπάρχουν ε, γεωργοί οι οποίοι έρχονται από τις άλλες χώρες και οι οποίοι ανακατεύονται στα πόδια μου λέει ο μιλητής και, και ε, καλλιεργούν το δικό μου έδαφος και αναγκάστηκα όχι μονάχα να τους μιλήσω αλλά και να τους δώσω και κάποιες συμβουλές και μπορώ να πω με μεγάλη χαρά και ευτυχία ότι παρά τις συμβουλές που τους έδωσα απέτυχαν. Πώς είναι δυνατόν να καινοτομήσει κανείς, πώς περιμένετε να καινοτομήσει κανείς εάν ε, οι καινοτόμοι τελικά φεύγουν και, παίρνουν τις ιδέες τους αλλού. Ο Σικυρέσκη και μετά ο ε, Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Υποστηρίζω την ιδέα του να συζητήσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων και της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος πυλώνας ε, θα συνεισφέρει ή συνεισφέρει ακριβώς για να αλλάξουμε την πραγματικότητα όπως έχει σήμερα. Έχει νόημα αυτό. Το νόημα, η ερώτηση ήταν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν αυτές οι προσαρμογές ε, και κατευθύνσεις. Γνωρίζουμε τα σχετικά ο πρώτος πυλώνας είναι για γενικές δράσεις και δραστηριότητες και δεν είναι αρκετά εξειδικευμένος και στοχοθετημένος από την ίδια του τη φύση. Γνωρίζουμε ότι η κερδοφορία όσον αφορά την αηφορία των μέτρων στην ανάπτυξη της υπαίθρου είναι ένας από τους στόχους για την ε, ανάπτυξη με τα μέτρα για τη γεωργία. Αυτό είναι το ερώτημα. Τίθεται ακριβώς αυτό το ερώτημα. Είναι εποφελής ε, σε σχέση με το στόχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας αυτό που είναι και ο τίτλος εξάλλου της μελέτης η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα βοηθούν όλα αυτά τα θέματα σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας ε, περιβαλλοντικής προστασίας όταν έχουμε ζητήματα καινοτομίας ε, ανταγωνιστικότητας τα καταφέρνουμε αυτά να υπάρξει μια ας το πω έτσι ένας συγκερασμός είναι μια απόλυτα νέα καινοτόμα δράση όταν είπε ο Επίτροπος Φίσλερ για το πώς ε, προχωρούσαν τα πράγματα και προς ποια κατεύθυνση έβαιναν και για τις κινήσεις όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, το ερώτημα είναι αυτή η στρατηγική αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 ή όχι. Ή μήπως δεν έχουμε καν στρατηγική σφαιρικά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και βρισκόμαστε σε κρίση και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την οικονομική κρίση συνολικά. Τα μέσα και τα εργαλεία στον πυλώνα 2 θα έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματικά. Αν λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση, τότε γιατί οι γεωργοί στην Ευρώπη δεν επιθυμούν να προσεγγίσουν τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα και να ενταχθούν σε αυτόν. Για τον πυλώνα ακριβώς δύο, είναι ακριβώς θα έλεγα δεν, δεν ευθυγραμμίζεται με εκείνο το οποίο θα έπρεπε να είναι. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με την γεωργία και για να προστατεύεται επίσης όμως και το περιβάλλον. Η ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου, των χώρων της υπαίθρου, φαίνεται όμως ότι απουσιάζει μέσα σε αυτό το ψηφιδωτό που πρέπει να συμπληρώσουμε με μέτρα και πρωτοβουλίες και η πολιτική για τη συνοχή είναι ένας επιπλέον συντελεστής. Φαίνεται ότι έχουμε πολιτικές για την υποστήριξη των αστικών και περιαστικών χώρων και παρότι δεν είναι αυτό εκείνο το οποίο ε, είναι ε, το κυριότερο για το οποίο πρέπει να κάνουμε λόγο για την ανάπτυξη της υπαίθρου, κάνουμε λόγο γενικά για την, την ε, βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Χάνουμε όμως τα θέματα για την γεωργία. Δεν μπορεί να αυτορυθμίζονται τα θέματα της γεωργίας οι γεωργοί να αυτορυθμίζουν τις δράσεις τους. Εξαρτώνται από εξωτερικούς συντελέστες και παράγοντες όπως το κλίμα, τις καιρικέ συνθήκες. Εμείς σχεδιάζουμε τώρα πράγματα για χρηματοοικονομικές αγορές και Κενώνεται έτσι περιεχομένου ο κανονισμός, ε, τα μέτρα για την ε, διαρθρωμένη γεωργία και για την ρύθμιση των αγορών και εδώ σε σχέση με θέματα του που ε, βλέπουμε ότι αγνοούνται αυτά τα σημεία και αυτά από τις, το πλαίσιο των προτάσεων. Και τέλος για το leader, για σχετικές δράσεις από πλευράς του leader και που αξιολογήθηκαν με διάφορους, διάφορους τρόπους. Πρέπει να μπορέσουμε να δούμε ότι κάποιοι ενεργοί πολίτες ε, χρησιμοποιούσαν το Λίντερ ιδιωτελώς <laughs> Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί όταν αξιολογούμε τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα δράσεων υπό το πλαίσιο του προγραμμάτος Leader. Και τέλος πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χρηματοοικονομικών μέσων που θα υποστήριζαν ή θα στοχοθετούσαν ποσοστά όσον αφορά δάνεια και πιστώσεις που θα ε, ε, ε, επιτρέπαμε να διατεθούν ώστε να υπάρξει πραγματικότητα θετική ε, ας το πω έτσι επίπτωση στην ανάπτυξη και να υπάρξει ευθύνη που θα επομίζονται όταν δέχονται κάποιες, κάποιες τέτοιες πιστώσεις και δάνεια. Αυτό ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κλάση. Ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε. Έχουμε εδώ έναν φιλόδοξο τίτλο. Αν ακούσει κανείς αυτόν τον τίτλο, πώς μπορούμε να πετύχουμε την ε, αηφορία και τη βιωσιμότητα στην γεωργία και για την ανταγωνιστικότητα. Με κάποιες τέτοιες στερεότυπες έννοιες κάνουμε εδώ επανειλημμένα χρήση. Αηφορία, ανταγωνιστικότητα, βέλτιστη χρήση και μετά από τα όσα είπε μόλις ο συνάδελφος Σικιόρσκι πιο πριν, και συγκρίνουμε το τι γίνεται και σε άλλες παρεμβάσεις διαπίστωσα ότι γίνεται αυτό, καθένας έχει τις δικές του σκέψεις και ιδέες όταν γίνεται λόγος για ηφορία και όταν προβληματιζόμαστε ο καθένας ε, για θέματα ηφορίας και βιώσιμης ανταγωνιστικότητας ή βιωσιμότητας. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη για την αηφορία και την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος για παράδειγμα. Σε σχέση με το περιβάλλον συνδέουν κάποιοι αυτή την έννοια. Και εδώ αυτό προκάλεσε κάποιες αντιστάσεις. Αηφορία ή βιωσιμότητα είναι κάτι παραπάνω από το περιβάλλον. Όχι μόνο η αηφορία και η βιωσιμότητα για τις θέσεις απασχόλησης που έχουμε επίσης για την αηφορία ή βιωσιμότητα των εισοδημάτων σε πολύ σημαντικά επαγγέλματα για να μπορούμε να έχουμε και υγιή υγειονομικά υγειονομικά και την πτυχή της ασφάλειας τρόφιμα. Όλα αυτά λοιπόν βιωσιμότητα, αηφορία, μπορούν έτσι να καθοριστούν μέσα σε αυτή την έννοια. Και η φορεία ή βιωσιμότητα ερμηνεύεται πάλι και διαφορετικά από τους πιο πολλούς. Αν δούμε αυτή τη μελέτη τώρα που έχουμε μπροστά μας, φυσικά πολλοί ευφιέστατοι άνθρωποι προβληματίστηκαν για αυτά τα θέματα και διατύπωσαν προτάσεις. Τότε επιτρέψτε μου και μένα να ρωτήσω, στο συνολικό αυτό φάσμα για τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις, μέσα στις μεταρρυθμίσεις για τη Γεωργία και στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα, βρήκατε κάτι υπό την έννοια αυτή και αυτή η έννοια τώρα είναι καινούρια θα έλεγα όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά και την πολιτική για την ανάπτυξη. Κάνουμε ξαφνικά λόγο για βλαπτικές, επιζήμιες στο περιβάλλον επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει πραγματικά κάτι τέτοιο, επιζήμιες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις και αν ναι, πώς μπορεί να οριστεί αυτό, να προσδιοριστεί. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν τέτοιες ε, στο περιβάλλον αρνητικές επιζήμιες τέτοιες επιδοτήσεις, αλλά υπάρχουν εδώ οι επαΐοντες που μπορούν ίσως να συνεισφέρουν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα πιο επιστημονικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάριαντ και μετά ο Κάπουλα Σάντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και για την παρουσίαση. Νομίζω ότι ο κύριος Κάς αναφέρθηκε σε ορισμένα από τα σημεία τα οποία ήθελα να, αναφέρω. Παρ' όλα αυτά, να ρωτήσω, ποια είναι η διασύνδεση ανάμεσα στο εισόδημα και την καινοτομία. Γιατί αν, υπάρχει σωστό, ε, αν υπήρχε μάλλον το σωστό εισόδημα στην ε, ε, Γεωργία, δεν θα μιλούσαμε για αυτά τα μεγάλα προγράμματα καινοτομίας. Επίσης έχουμε κάποιους αυστηρούς ε, ε, κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης. Μπορεί κανείς να συμφωνήσει, να διαφωνήσει σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων σε σχέση με την βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Επίσης στο σημείο 11 μιλάτε για αναδιανομή ε, του πυλώνα 1 όπου το κυρίαρχο στοιχείο είναι η ε, δικαιοσύνη και λέτε και η ίδια ότι εκεί χρειάζονται αντικειμενικά κριτήρια. Έχετε κάποια τέτοια αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να εφαρμοστούν εκεί. Χαίρομαι που έχουμε τη συζήτηση αυτή γιατί είναι πολύ ουσιαστική, αλλά όσον αφορά συγκεκριμένα πρακτικά αποτελέσματα, πιστεύω ότι κάποιες από τις ιδέες που περιέχονται εδώ θα αφορούσαν καλύτερα το επόμενο βήμα και όχι το βήμα που έχουμε τώρα μπροστά μας. Ας πούμε στη σελίδα 46 της έκθεσης λέμε ότι χρησιμοποιούμε λιγότερα ε, λιγότερα ε, ζυζανιοκτώνα λοιπά Αλλά αυτό είναι ας πούμε το βιώσιμο. Επίσης ε, μιλάμε για μόνο για την εσωτερική αγορά ή γενικά για την παγκόσμια αγορά, γιατί βλέπουμε ότι η παραγωγή μας χάνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τελευταία παρατήρησή μου που ελπίζω ότι θα διατυπωθεί σωστά σαν ερώτηση είναι η εξής. Βεβαίως Εάν ξεκινούσαμε τώρα να κάνουμε μια πολιτική για τη γεωργία, δεν θα, είμαστε, δεν θα ξεκινούσαμε από αυτό το σημείο, όμως εδώ είμαστε. Και δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τα πάντα. Αυτό είναι ένας κίνδυνος, το να καταστρέψουμε τα ε, ήδη υπάρχοντα. Δηλαδή να αυξηθεί τόσο η γραφειοκρατία και η περιπλοκότητα που να καταστραφούν τα πάντα. Συμφωνώ με τα προγράμματα του πυλώνα 2, μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά, αλλά όσο πιο στοχευμένος γίνεσαι, όσο πιο συγκεκριμένος γίνεσαι, τόσο πιο περίπλοκος γίνεσαι. Άρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Ευχαριστώ. Λουίς Κάπουλα Σάντος και θα κλείσει ο Κόσιγκερ. Ελίζαμπεθ. Όχι, συγγνώμη, θα κλείσει η Ελίζαμπεθ Κόσιγκερ, ο κύριος ε, Κάμπος. Ήθελα μόνο να ευχαριστήσω για αυτή τη μελέτη Κρίμα που δεν μπόρεσα να το διαβάσω αυτό πιο πριν ως έγγραφο, γιατί είναι ένα έγγραφο το οποίο απαιτεί πολύ προσεκτική ανάγνωση. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα αυτά, θα είμαι πραγματικά πολύ φιλομαθής για να δω πού καταλήγει και σε τι θεμελιώνονται τα συμπεράσματα τα οποία μας έχουν υποβληθεί, διότι πραγματικά είναι πραγματικά θα έλεγα συγκλονιστικά. Εμείς αναζητούμε μια μεταρρύθμιση που θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ταυτόχρονα με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας σε ένα πλαίσιο αηφορίας. Και εδώ αμφισβητεί, ας το πω έτσι, θέτει ενώπιόν μας η έκθεση με σαφήνεια ότι τα μέτρα τα οποία προετοιμάζουμε μπορούν να ε, έχουν επίπτωση σε αυτούς τους στόχους. Και ε, τοποθετείται σαφώς ε, υπέρ της, ε, του δεύτερου πυλώνα στα μέτρα η συγγήτρια μετά από μια πρώτη ανάγνωση που έκανα και λέει ότι η ΚΑΠ πρέπει περισσότερο να προσεγγίζει μια αναθεώρηση μέσα στον δεύτερο πυλώνα και όχι τόσο στην εστίαση στον πρώτο πυλώνα και προτείνει ο δεύτερος πυλώνας να έχει τουλάχιστον 40% δεν το κατανοώ απόλυτα. Πώς βρίσκεται αυτό το κατόφλι, πώς καθορίζεται, πώς μπορεί αυτό το κατόφλι να συνεισφέρει για να επιτύχουμε αυτού του είδους τους στόχους αποτελεσματικά. Εν πάση περιπτώσει, τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς είμαι εισηγητής για τις άμεσες πληρωμές, για τον πρώτο πυλώνα και την ανάπτυξη των μέτρων του δεύτερου πυλώνα, προσπάθησα και ε, εδώ και σε σχέση και με την ε, ολοκλήρωση αυτών των ε, εκθέσεων που σύντομα θα είναι μέσα οι εκθέσεις αυτές η μεγάλη προσπάθεια που έκανα είναι να έχω ένα συνεκτικό πλαίσιο και ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τους δύο πυλώνες ώστε το σύνολο αυτών των μέτρων να μπορέσει να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε ενώπιόν μας. Επαναλαμβάνω, μια ανταγωνιστική γεωργία αλλά προφανώς μέσα στο πλαίσιο του σεβασμού του περιβάλλοντος και της αηφορίας, της σταθερής αηφορίας αυτό σε σχέση με, αυτή τη, με αυτό το έγγραφο. Το θεωρώ χρήσιμο βέβαια, διότι θα μας βοηθήσει κάποια θέματα να τα αποσαφηνίσουμε και να επανορθώσουμε ή να διορθώσουμε κάποιες τοποθετήσεις κάποιων εκθέσεων στα θέματα υποσυζήτηση και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω για τη σύνταξη αυτής της μελέτης την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Ελίζαμπετ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση της μελέτης. Πιστεύω ότι πολλά ήδη προαναφέρθηκαν Κυρίως ε, και όσον αφορά αυτά τα θέματα τα οποία προαναφέρθηκαν συμμερίζομαι την άποψη για τη σπουδαιότητα και για το δυναμικό που υπάρχει στον δεύτερο πυλώνα που πρέπει να προσέξουμε. Το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου να έχουμε την μέγιστη ελαστικότητα στα κράτη-μέλη που θα διασφαλίζεται για τα κράτη-μέλη και κυρίως να έχουμε ένα σύστημα κινήτρων που θα χρησιμοποιούμε και θα πρέπει βλέποντας ποια κράτη είναι επιτυχή στον τομέα της ανάπτυξης υπαίθρου, π.χ. χώρες που πραγματικά ωφέλησαν με τα μέτρα τους τους γεωργούς και πρόσφεραν μέτρα για το περιβάλλον και το χώρο της υπαίθρου, έτσι πρέπει να δούμε ότι είναι αποτελεσματικά και λειτουργούν. Για μένα υπάρχει όμως μια αντίφαση όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής. Γιατί η Επιτροπή τον τομέα της συνάρτησης με τον τουρισμό για τη γεωργία τον έχει αφαιρέσει, τον θέτει εκτός ε, πλαισίου και ιδιαίτερα όσον αφορά εκμεταλλεύσεις, όσον αφορά οικογενειακές εκμεταλλεύσεις γεωργών ε, που δεν προσέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ίσως θα έπρεπε να δει τέτοιε δυνατότητες η Επιτροπή και να υποβάλει προτάσεις ιδιαίτερα για την αηφορία αφενός και για την καινοτομία, καινοτόμες δράσεις και επενδύσεις αφετέρου. Και σίγουρα αυτό θα μπορέσει να συνεισφέρει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο μέλλον. Διότι ακόμα και σε εντατικέ εκτάξει καλλιέργεια θα μπορούσαμε τέτοιε εναλλακτικέ λύσει να τι προτείνουμε. Και για τι επενδύσει όσον αφορά την αηφορία του πιο μακροπρόθεσμα και σε αυτό τον τομέα, κανένα δεν μπορεί να έχει αντίρρηση. Απ' την άλλη πλευρά όμω θα πρέπει να σκεφτούμε ακριβώ ποιοι συντελεστέ και ποιοι δείκτε θα είναι αυτοί που θα λαμβάνονται υπόψη ακριβώ στον τομέα τη γεωργία υπάρχει μια περιφέρεια ή περιοχή που να εξισώνεται και να γίνεται ταυτόσιμη με μια άλλη όσον αφορά τι ανάγκες της ή όπως το ίδιο σημαίνει και με μια εκμετάλλευση και μια άλλη. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές και διαφοροποιημένα πρέπει να λυθούν αυτά τα στοιχεία υπόψη για την αποτελεσματικότητά τους. Όσα ισχύουν για τη μία περιφέρεια δεν μπορούν να ισχύουν για άλλη περιφέρεια ή άλλη εκμετάλλευση ισοπεδωτικά. Και όσον αφορά τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν συμφωνώ με τους συναδέφους. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η συμβουλευτική δραστηριότητα μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις. Και εδώ πάλι υπάρχουν οι πιο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ένα άλλο σημείο και εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι γι' αυτό, γιατί επανειλημμένα σε όλους τους τομείς αυτό προτείνεται ή αναφέρεται όταν αναφέρονται οι δείκτες ή ενδείκτες η γραφειοκρατική, η γραφειοκρατία είναι ένα απόλυτο πρόσκομα, ένα εμπόδιο για τις επενδύσεις. Δεν χρειάζεται αυτό να ε, το τονίσουμε γιατί η σημασία του είναι θα έλεγα κάθετη. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη και μια συγκεκριμένη ερώτηση, μια και δεν αναφέρθηκε αυτό στην έκθεση. Τι θα γίνει με τις περικοπές όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Περικοπές ε, όσον αφορά την αηφορία και την βιώσιμη ανταγωνιστικότητα για τις επενδύσεις. Έχουμε κάποια ποσά που ακούγονται, κάποια ποσοστά για περικοπές. Ακούγονται 100 δισεκατομμύρια λέει ευρώ που θα εξοικονομηθούν με περικοπές. Τι θα γίνει για την ανάπτυξη συμπέθρου και με τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα για την πολιτική για την γεωργία 30 δις ευρώ θα ήταν λέει αυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε ποιες άμεσες επιπτώσεις θα υπάρξουν σε σχέση με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη μέσω τέτοιων μέτρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ελίζαμπετ, σας ευχαριστώ όλους. Ξαναδίνω το λόγο στους εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν στις ερωτήσεις και εγώ θα ήθελα μαζί όπως και οι συνάδελφοι να ευχαριστήσω τους καθηγητές για την παρουσίασή τους. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι και ελπίζω ότι οι συγητές μας θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις προτάσεις της Κομισιόν, περιλαμβάνοντας και χμές από τις τοποθετήσεις των εμπειρογνωμόνων μας, για να μπορέσουμε να έχουμε μια γεωργία πιο ανταγωνιστική, πιο αποτελεσματική που δεν θα την εμποδίζουμε με περαιτέρω γραφειοκρατία. Ο, κύριος, ο καθηγητής Blackwell θα απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους ε, βουλευτές ε, για αυτές τις έξι σελίδες σημειώσεων που πήρα σχετικά με τις ε, ερωτήσεις. Αλλά βεβαίως και αν κάτι δεν απαντηθεί μπορείτε να έρθετε σε επαφή δημιουργός μαζί μας. Θέλω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και μετά να αποσαφηνίσω τα όσα θέλαμε να σας πούμε εδώ έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε στις ενέργειες που θα ακολουθήσετε όσον αφορά την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Είχαμε, ακούσαμε 12 ε, ερωτήσεις και διεπίστωσα αμέσως ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν αναφέραμε. Το ένα ας πούμε ήταν η συγχρηματοδότηση. Ούτε η Κομισιόν δεν θίγει το θέμα αυτό γιατί είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Παρόλα αυτά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διότι στην ουσία έχουμε δώσει το μήνυμα ότι πρέπει να δοθεί έμφαση ε, σε αυτά τα οποία παραδοσιακά μπαίνουν ε, στον πυλώνα 2, αλλά από τη στιγμή που στον πυλώνα 2 υπάρχει συγχρηματοδότηση υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν έχουν χρήματα τα κράτη-μέλη για, επιπλέον χρηματοδότηση. Η προσωπική μου γνώση, ε, γνώμη είναι ότι θα πρέπει εδώ να κάνει πίσω η συγχρηματοδότηση και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και από την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο όντω δεν αναφέραμε και καλά έκαναν οι βουλευτές και το έθιξαν. Τουλάχιστον δύο ε, βουλευτές αναφέρθηκαν στην ασφάλεια και πολύ σωστά το αναφερθήκατε στην ασφάλεια. Είναι ζωτικής ε, σημασίας ε, σημείο για την διατροφική αλυσίδα ε, και βεβαίως ε, δεν νοείται ΚΑΠ χωρίς προμετωπίδα την, τα ασφαλή τρόφιμα. Είναι όμως ένα σημείο το οποίο δεν πολύ προσέξαμε και οπωσδήποτε χρήζει συζητήσεως. Ε, η άποψή μας ε, είναι ταυτόσιμη με το Κοινοβουλίου, δηλαδή ότι θα πρέπει η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να βοηθήσει ε, και τους χρήστες που δεν είναι γεωργοί και που μπορεί να βοηθήσει την Ήπεθρο να γίνει μια βιώσιμα αναπτυγμένη περιοχή με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχουν, θα υπάρχουν άτομα που δεν θα είναι ε, κατά κύριο λόγο ε, γεωργοί, αλλά θα πουλούν τα ε, θα πουλούν τα γεωργικά προϊόντα και έτσι ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους και έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα υγιές αγροτικό και ε, πλαίσιο για ένα πλαίσιο υπαίθρου υγιέστερο. Υπάρχει κάποιος στην Ευρώπη άραγε που να μην υποστηρίζει ότι θα πρέπει η Γεωργία να είναι ανταγωνιστική ή τέλος πάντων να γίνει πιο ανταγωνιστική από ό,τι είναι τώρα και ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι βιώσιμη ε, με την έννοια ότι ε, δεν θα μειώνει το φυσικό κεφάλαιο, δεν θα ε, λερώνει και δεν θα μολύνει το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα και ότι τέλος πάντων οι Γεωργοί μεταξύ άλλων θα παράγουν και θα παρέχουν και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Φαντάζομαι φαντάζομαι πως δεν υπάρχει ούτε ένας. Το ζήτημα είναι ποια θα είναι η ισορροπία για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη ε, το που βρισκόμαστε τώρα, στην επόμενη εκστρατεία της ε, ΚΑΠ θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν την εστίαση στην ε, βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, στην ασφάλεια ή θα πρέπει απλώς να προχωρήσουμε έτσι ώστε να δούμε πώς είναι δυνατόν να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα αλλά προσπαθώντας κυρίως να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα. And the Commission is we've got to do both. Και για να μπερδέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο για τη βιωσιμότητα στον ε, πυλώνα 1, εκεί δηλαδή που εντάσσεται το πρασίνισμα κυρίως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τον τρόπο αυτό. Δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πέραν τούτου όμως, στην έκθεσή μας κυρίαρχο στοιχείο είναι το εξής. Εάν ε, δείτε την, ε, τα μεταποιητικά, τα μεταρρυθμιστικά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν ε, την γεωργία να προσαρμοστούν. Τα περισσότερα μέτρα βρίσκονται στον πυλώνα 2, δηλαδή εξυγχρονισμό της παραγωγής και της διεμπόρευσης, βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, συνεργασία βελτίωση της συνεργασίας, η ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, αυτές όπου τα στοιχεία της φύσης είναι πιο ε, σκληρά, ε, προώθηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων κτλ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες εστιάζονται και στην βιωσιμότητα και στην ανταγωνιστικότητα, στην ουσία, στο, στο μεγάλο τους μέρος βρίσκονται στον πυλώνα 2 και το πρόβλημα είναι ότι δεν, θέλει, δεν υπάρχει βούληση διεύρυνσης του πυλώνα 2 ή ε, μετακύλησης κάποιων από τα στοιχεία στον πυλώνα 1. Ζητούμε από τους ε, γεωργούς να προσέξουν περισσότερο το περιβάλλον, να, να προσέξουν περισσότερο τις γεωργικές τους πρακτικές, αλλά τίποτα περισσότερο. Δεν τους βοηθούμε παραπάνω και επομένως ε, η Επιτροπή Γεωργίας εδώ ε, πρέπει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να καθοδηγήσει προς το σωστό μέρος, ε, προς, τι προς τις σωστές διαδικασίες και τη σωστή επιχειρηματολογία την συζήτηση, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούν να ενδυναμωθούν οι αντιπροτάσεις αυτές, οι counter proposals. Και θα ήθελα να πω και δύο λόγια. Το θέμα του προπολογισμού είναι σημαντικό. Οι φίλοι της Ευρωπαϊκής ε, Γεωργίας ε, ζητούν βεβαίως ε, ισχυρό προϋπολογισμό και πρέπει να ζητούν ισχυρό προϋπολογισμό για την γεωργία γιατί διαφορετικά και στο σκέλος της βιωσιμότητας και στο σκέλος της ανταγωνιστικότητας υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας. Και θα, θα περάσω τώρα το λόγο στην Τζάνετ. Πολύ σύντομα να αναφέρω κάποιες λεπτομέρειες ε, που ακούστηκαν σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα τα οποία θέσατε και για τα οποία σας ευχαριστώ. Ε, αναφερθήκατε στην επίστοση, σαν, ε, την πίστη μάλλον, ε, σαν ε, μοχλό ανάπτυξης των περιοχών. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε έτσι πιο εφάνταστους τρόπους τοπικής άντλησης ε, χρημάτων ε, και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει πάρα πολύ τους γεωργούς στις περιφέρειες κυρίως αυτές, στις περιοχές κυρίως αυτές όπου δύσκολα μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια οι γεωργοί. Τώρα, το θέμα του, της διαχείρισης κινδύνου, risk management και πώς λειτουργούν ας πούμε τα μέτρα αυτά στην Βόρεια Ιταλία. Ε, εκεί ε, υπάρχει γενική αίσθηση ότι δεν είναι η σωστή θέση αυτής της διαχείρισης κινδύνου στον πυλώνα 2 γιατί ούτως ή άλλως ε, είναι πιο λογικό σε πολλές περιπτώσεις ε, ε, αυτή η διαχείριση να γίνεται σε επικεντρωμένο εθνικό επίπεδο και όχι σε περιφερειακό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τα σημεία σχετικά με την συμβουλευτική και τι εννοούμε όταν λέμε συμβουλευτική παροχή συμβουλών, όταν δίνει συμβουλές ε, βοηθάς ε, κάποιον ε, να πάρει σωστές αποφάσεις. Δεν του υποβάλλεις αποφάσεις. Είναι μια κινητροδότηση κατά κάποιο τρόπο. Ε, έτσι ώστε να βοηθήσεις ε, τους ε, ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν, να ξεπεράσουν κάποια δυσκολία εν προκειμένου παροχή συμβουλών έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους γεωργούς να καταλάβουν καλύτερα και να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Ρωτήσατε πιο στοχευμένη βοήθεια σημαίνει περισσότερο κόστος και μεγαλύτερη γραφειοκρατία πρόβλημα είναι ότι εδώ κοιτάμε πάντα την αρχική φάση, αυτή τη startup phase. Αλλά εάν θέλετε πραγματικά να δημιουργήσετε, ε, να οικοδομήσετε διατομεακές εταιρικέ σχέσεις, ε, τότε θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν οι μεν τους δε. Αν δεν υπάρχει άλλη κατανόηση, αν δεν δοθεί κάποιος χρόνος ε, για πραγματικό διάλογο, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην επόμενη φάση. Ε, βλέπουμε ότι προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, ε, εκεί όπου έχει υπάρξει διάλογος, εκεί που ο κόσμος έχει αρχίσει να κατανοεί ο ένας τον άλλον, ε, προχωράνε χωρίς ιδιαίτερο λειτουργικό κόστος. Πιστεύω ότι εξ αρχής θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, να διαπλέξουμε τέτοιες σχέσεις έτσι ώστε να, να μειωθεί το κόστος σιγά σιγά. Ε, και ξέρετε μπορεί αφιψηλού μερικά πράγματα να φαίνονται πολύ καλά αλλά εάν κατεβεί κανείς σε τοπικό επίπεδο βλέπει ότι ε, δεν υπάρχει καμία διασύνδεση μεταξύ των στοιχείων των ανθρώπων και τα λοιπά και των προσπαθειών και επομένως τίποτα δεν λειτουργεί. Ένα κουβάρι γίνονται όλα. Ε, και επομένως δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, το αντίθετο μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και πάλι τους εμπειρογνώμονές μας. Παρακαλώ τώρα τον ε, Διευθυντή, τον κύριο ε, Πλέβα, αν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω κάτι ότι η ανταγωνιστικότητα, η αηφορία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας είναι ένας από τους κύριους πυρήνες της κοινή αγροτικής πολιτικής και η καινοτομία πραγματικά είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ακούσαμε την παρουσίαση και διαβάσαμε και το έγγραφο με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά και ακούσαμε και διαβάσαμε και βλέπουμε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, τοποθετήσεις, ιδέες για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠΑ αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο έντονων σε βάθος διαπραγματεύσεων και στην Ευρωβουλή αλλά και στο Συμβούλιο. Και αυτό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυσχεραίνει τα πράγματα να συζητηθούν τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης σε αυτή τη φάση, υπό αυτή τη συγκυρία. Διότι άμεσα αναφέρεται η μελέτη στις προτάσεις της μεταρρύθμισης και οι προτάσεις της μεταρρύθμισης ήταν αντικείμενο σε βάθος ανάλυσης επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Impact Assessment, μελέτη επιπτώσεων, καλύπτει επίσης το θέμα της αηφορίας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας. Εν τούτης, ως πρώτη αντίδραση, θα ήθελα να τονίσω κάτι. Να τονίσω ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια ανάγκη να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα περισσότερο. Αποσαφήνιση, διευκρίνηση λοιπόν περισσότερο για τον ρόλο της εταιρική σχέσης για την καινοτομία μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Υπάρχει η προθυμία να υπάρξουν αυτές οι αποσαφηνίσεις έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως είναι αναγκαίο και σε σχέση και με τους συντάκτες της μελέτες από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δευθύντα Πάμε στο σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Αλλαγή του κανονισμού 1234 για την υποστήριξη ε, στους αμπελιοκαλλιεργητές. Ο Χέρμπερ Ντόρφμαν έχει το λόγο. Ο εισηγητής μας συνεργάστηκε στενά και με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν για να βρει μια κατάλληλη λύση για το θέμα που να εγγυάται την απαραίτητη ευελιξία για τις μελλοντικές πολιτικές αποφάσεις στον αμπελοϊνικό τομέα. Παρακαλώ, Χέρμπερτ, έχει το λόγο και εξήγησέ μας αναλυτικά το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, αυτή η έκθεση είναι τμήμα του συνολικού πακέτου μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, κοινή αγροτικής πολιτικής. Και επίσης, εκείνη από τη διαπίστωση ότι θεωρεί ότι το, τα υπόλοιπα μέτρα του πακέτου για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ιδιαίτερα για τον πρώτο πυλώνα, θα λειτουργήσουν όπως έχει σχεδιαστεί τώρα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για όλες τις, γεω, τις ε, ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μεταποίησή τους να υπάρχουν απαιτήσει πληρωμών στον πρώτο πυλώνα όταν τίθενται αυτές. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν τώρα όταν έχουμε τους αμπελουργούς και εινοποιούς θα έχουν τέτοιες απαιτήσει και όταν θα τις έχουν από πού θα προέρθουν αυτά τα κονδύλια και ουσιαστικά για τον σήμερα διαθέσιμο προϋπολογισμό για τον πρώτο πυλόν από το Single Payment Scheme έρχονται αυτά τα κονδύλια. Όμως θα συμβεί το εξή. Για τον τομέα τον εινοποιητικό μέσω της ρύθμισης ε, για τον κανονισμό για την αγορά που μεταρρυθμίστηκε πρόσφατα έχει ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό που στους εθνικούς, στα εθνικά χαρτοφυλάκια National Envelopes διοργανώνεται στην κοινή οργάνωση αγοράς για την εινοποίηση και βρίσκει χρήση σε αυτά τα εθνικά χαρτοφυλάκια από πλευρά των κρατών μελών. Έτσι αποφασίζονται οι ενισχύσεις, τα κονδύλια που διατίθενται. Σε αυτή την έκθεση θα πρόκειται τώρα για το εξής, να έχουν την εναλλακτική λύση όχι υποχρεωτικά, αν θέλουν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν έτσι τα κράτη-μέλη, ένα μέρος ή το σύνολο του εθνικού χαρτοφυλακίου να μπορούν να το διαθέτουν, να το χρησιμοποιούν, ώστε να καλύπτονται οι άμεσες πληρωμές στον τομέα των εινοποιητικό, στον πρώτο πυλώνα ή έτσι να χρηματοδοτούνται. Με άλλα λόγια μπορούν ένα μέρο ή το σύνολο του Εθνικού Χαρτοφυλακίου National Envelope να το εντάσσουν σε αυτόν τον προπολογισμό για τι άμεσε πληρωμές για τον πρώτο πυλώνα και έτσι να γίνονται τα εμβάσματα και οι πληρωμέ, ώστε οι πρόσθετε δαπάνε που θα απορρέουν σε σχέση με την εινοποιία για τι εκτάσει ε, και για τις επιδοτήσιμες εκτάσεις του πρώτου πυλώνα έτσι να καλύπτονται και οι δαπάνες έτσι στον πρώτο πυλώνα θα μπορούν να καλύπτονται σε αυτό το πλαίσιο. Και σε σύμφωνη γνώμη πάντα και συντονισμό, τουλάχιστον αυτό προβλεπόταν στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν αν θα το κάνουν αυτό ή όχι, στη δική τους διακριτική ευχέρεια. Θα πρέπει να μπορεί αυτό έτσι να λειτουργήσει το 2012 με αυτόν τον τρόπο, ώστε το 2014 αν χρειαστεί να έχουμε μεταθέσεις κονδυλίων, μεταφορές κονδυλίων όπου είναι αναγκαίο. Και σε σύμφωνη γνώμη με το Συμβούλιο, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο, βρήκαμε μια μεταβατική προσωρινή λύση ως εξή δηλαδή. Μέσα στο ίδιο το πλαίσιο του 2012 θα πρέπει μέχρι την εκνοή του 2012 να αποφασίσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη αν για το 2014 ή αποκλειστικά για το 2014 τμήματα ή το συνολικό χαρτοφυλάκιο ως άμεσες πληρωμές θα το διαθέτουν ή όχι. Είναι μια εφάπαξ μία και μόνο απόφαση που θα ληφθεί για αυτή την ε, λειτουργία και αν θέλουν να επανέλθουν μετά το 2014 στο Εθνικό Χαρτοφυλάκιο, αν το επιθυμούν, μπορούν τότε να το κάνουν. Μέσα όμως το ίδιο το 2013 το ίδιο θα πρέπει να αποφασίσουν τελεσίδικα και καθοριστικά τα κράτη-μέλη, αν επιθυμούν να γίνουν αυτές οι μεταφορές. Και έτσι από το 2015 εφ' εξής, με ένα αξισίο το 2015, αυτές ε, οι μεταφορές ε, οι πληρωμές αυτές δεν θα μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ μέσα στο πλαίσιο ή να καταργηθούν ε, διότι θα έχουν ενταχθεί μέσα στις ε, απαιτήσει όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα και δεν θα μπορούν να αποσυνδεθούν όσον αφορά το single payment scheme από αυτό το πλαίσιο. Κατά τούτο υπάρχει λοιπόν συνεννόηση με το Συμβούλιο να λειτουργήσουν έτσι τα πράγματα. Όλες οι άλλες τροποποιήσεις ε, και τα λοιπά έχουν ε, μικρότερη σημασία, είναι πιο εξειδικευμένες. Έχω καταθέσει μια πρόσθετη τροπολογία όπου προτείνω να υπάρχει δυνατότητα που θα παρέχεται στα κράτη-μέλη να αφήσουν τα πράγματα όσον αφορά την ε, χρηματοοικονομική επιβάρυνσή τους όσα έχουν, δηλαδή η οποία να βγει από το Single Payments ε, Scheme, να μην είναι δηλαδή υποχρεωτικός ο πρώτος πυλώνας, να παραμένουν στο εθνικό χαρτοφυλάκιο για την εινοποιία όπως προβλέπεται και σήμερα και να διατηρηθεί αυτή, αυτό το πλαίσιο και για το μέλλον, να μην ενταχθεί στο Single Payments ε, Scheme. Αυτές είναι οι περισσότερες ε, οι καινοτομίες που υπάρχουν με λίγα λόγια συνοπτικά. Ευχαριστώ. Grazie, Ευχαριστώ Χέρμπερτ, ήσουν σαφέστατος. Τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση. Και θα δώσουμε και το... Εράντς Καρσία είναι η πρώτη που θέλει το λόγο. Και μετά ο Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα, σκληρό, αντιπαθητικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την προσπάθειά του. Ο εισηγητής έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν έχει δίκιο η Κομισιόν που θέλει να που θέλει να επιταχύνει τα πράγματα, διότι έχουμε χρόνο μπροστά μας. Έχει δίκιο η συγητής. Είναι βιαστική απόφαση και μπορούμε να αφήσουμε χρόνο στα κράτη-μέλη. Επίσης, δεν συμμερίζομαι όλη τη γνωμοδότηση του εισηγητή. Γιατί η απόφαση για την επιλεξικουμότητα στις πληρωμές της ΚΑΠ θα ληφθεί από τον κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές. Θα ήταν λοιπόν λογικό μέσα σε αυτό το πλαίσιο των αμέσων πληρωμών να, θεω... να υπολογιστεί και το πριμ για την <coughs> αμπελοϊνική έκταση. Χρόνο πρέπει να αφήσουμε, όπως λέει και ο εισηγητής. και να αναφερθούμε κατευθείαν στον Γενικό Κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές. Ευχαριστώ. Ο Λουίς Κάπουλα Σάντος και μετά η κυρία Λούλινγκ. Θα ήθελα απλά και μόνο να επιστήσω την προσοχή για την ανάγκη να συσχετήσουμε αυτή την έκθεση με την πρόταση για τις άμεσες πληρωμές. Εξάλλου όπως πιο πριν ανέφερε η συνάδελφός μας. Αλλά και να δούμε αν θα μπορούσαμε να έχουμε την τοποθέτηση μετά από την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή της ε, Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Διότι το ερώτημα που τίθεται είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας θέσει την ημερομηνία 2012 σε ένα κανονισμό που συζητούμε και έχοντας θέσει τον κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές ε, την δυνατότητα αυτοί οι γεωργοί να μπορούν ε, να έχουν αυτή την επιλογή μέχρι τη 15η Μαΐου 2014 θα υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος για αυτή την επιλογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μόνο για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού για το εθνικό χαρτοφυλάκιο και την μετέπειτα κατανομή το, για τους συνοποιούς όταν θα ενταθούν σε αυτό το καθεστώς. Χρειάζονται αυτές οι αποσαφηνήσεις για τον καλύτερο τρόπο, ας το πω έτσι, άρθρωσης αυτών των στοιχείων. Και νομίζω ότι αν μπορεί αυτό να γίνει σε μια μετάθεση χρονικού ορίου υστερότερα, ώστε όταν θα έχουμε για τον κανονισμό για τις ε, άμεσες πληρωμές, θα ήταν κάτι καλύτερο. Αντί να υποχρεώσουμε υποχρεώσουμε τους γεωργούς πιο πριν να υποχρεώνται να κάνουν μια ε, επιλογή από πλευράς των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λουίς. Η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον Herbert Dorfman, γιατί Είμαι κάπως μπερδεμένη και θέλω να ρωτήσω για να δω αν κατάλαβα καλά. Διότι άμα δει κανεί τις τροπολογίες και τις μελετήσει στα γαλλικά, είναι κάπως αστείο. Σαν να θέλαμε να αποκλείσουμε δηλαδή την αμπελουργία, την αμπελοκαλλιέργεια από τις επιλέξιμες ζώνες. Κατάλαβα καλά. ευχαριστώ για αυτόν τον συμβιβασμό ότι δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να αποφασίζουμε, δηλαδή... Θα πρέπει να ξέρουμε πόσα περιέχει ο χρηματοδοτικός φάκελος. Εμείς για το δικό μου κράτος πήραμε τον εθνικό φάκελο για την αμπελοκαλλιέργεια και δώσαμε κουπόνια ανεκτάριο. Και αυτό μοιράστηκε ανεκτάριο. Σήμερα μπορούμε εμείς να κρατήσουμε αυτό, το φάκελο και αυτό το σύστημα, αλλά αν κρατήσουμε αυτό το φάκελο και αυτό το σύστημα, δεν εντασσόμεθα στο single payment scheme. Αλλά αν ενταχθούμε όμως στο single payment scheme, είναι σαφές ότι θα πρέπει να μοιραστούμε με τους άλλους. Οπότε ο χρηματοδοτικός φάκελος θα μικρύνει. Κατάλαβα καλά. Αν λοιπόν ούτως έχουν τα πράγματα για μας, διότι οι δικοί μας ε, αμπελοκαλλιεργητές είναι πανευτυχείς με τα μέτρα που έχουμε. Πήραμε το φάκελο, πήραμε το ποσό, το διαιρέσαμε ανεκτάριο και δώσαμε μία ενιαίο πριμ. Λοιπόν, κατάλαβα καλά. Είναι αυτό το οποίο πιστεύει η διπλανή μου ότι το κείμενο της Κομισιόν θα επέτρεπε και την άλλη δυνατότητα, δηλαδή να παραμείνει η αμπελοκαλλιέργεια στις επιλέξιμες περιοχές. Δεν κατάλαβα. Θέλω να ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιλογής που θα κάνουμε. Και μετά εντάξει ο φάκελος, αλλά να ξέρουμε και τι θα περιέχει. Εάν εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τον εθνικό χρηματοδοτικό φάκελο, πρέπει να ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσό αν αποφασίσουμε να μην κρατήσουμε αυτόν το φάκελο και να πάμε στο σύστημα των ενιαίων πληρωμών, πάλι δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο φάκελος και πάλι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επίπτωση του μοιράσματο με, την υπόλοιπη, με, τους ε, με τις υπόλοιπες καλλιέργειες, δηλαδή τι θα πάρει η αμπελουργία έναντι των άλλων. Ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ, ο Σέρτζο Γκουτιέρες. Πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω και να εκφράσω τη συμφωνία μου με τον κύριο Ντόρφμαν. Πρόκειται για μια πολύ τεχνική έκθεση. Δεν έχει τίποτα το πολιτικό, ούτε καν το αγγίζει. Βέβαια, κατά βάθος, κατά βάθος υπήρχε ένα πολιτικό ζήτημα σχετικά δηλαδή με τις δημοσιονομικές προοπτικές που όπως είπε και η συνάδελφος ε, δεν προμηνύεται και καμία ε, κοντινή συμφωνία που να ικανοποιεί και αυτά που ζητάει το Κοινοβούλιο. Και αυτή η απόφαση των κρατών μελών που θα έπρεπε να μας πούνε αν θα περάσουν στο, στο υπερεθνικό σύστημα ή όχι έχει μεγάλη πολιτική συμμαχία. Τέλος πάντων, εμείς δεν ψάξαμε τα, ψηλά γράμματα του τεχνικού σκέλους ε, και βρήκαμε το πολιτικό σκέλος και το εστιάζουμε αρκετά καλά. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία τις προθεσμίες μέσα στις οποίες ε, κινούμεθα, τα συμφέροντα που προασπίζουμε σε αυτή την περίπτωση και πιστεύω ότι πρόκειται για μια κατάλληλη στρατηγική να ζητήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία και μέσα στο χρόνο που θα επιτρέψει το στο να υπερασπιστεί τους ε, αμπελουργούς. Έχουμε τις ίδιες αμφιβολίες με την κυρία Εράντσα για το θέμα της επιλέξιμης έκτασης. Θα καταθέσουμε μια τροπολογία σχετικά. Και επίσης εδώ που φτάσαμε ήταν επιτυχία να μην βάλουμε, να μην εισάγουμε στη συζήτηση και το δικαίωμα θήτευσης. Μπορέσαμε δηλαδή να περιχαρακώσουμε την ουσιαστική συζήτηση. Και συμφωνούμε με τον εισηγητή σε αυτά τα οποία μας είπε για την αμπελοκαλλιέργεια και φυσικά σε τελευταία ανάλυση και για, τον, για την πρόθεση του κρασιού. Ευχαριστώ Σέρτζο. Μάρτιν. Ναι, πολύ σύντομα, πολύ σύντομα μόνο για να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Αν κατάλαβα καλά, πρόκειται για το ότι ουσιαστικά στο τέλος θα έχουμε κάθε κράτος μέλος που θα μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι αποτελεσματικό για μια κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε αν είναι ή όχι. Όμως μετά από συζητήσεις με ενώσεις παραγωγών εινοποιητών στη Γερμανία, οι εινοποιοί οι ίδιοι θα ήθελαν να έχουν το σύστημα πληρωμών με εκείνο το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή στην Γερμανία και που είναι ικανοποιημένοι με αυτό και με τη δομή των μικρών επιχειρήσεων, εινοποιητικών επιχειρήσεων δεν είναι αποφασιστική σημασία αν έχει κανείς 5, 6, 10 εκτάρια ή κατά μέγιστον αν θα παίρνει το πριμ για αυτή την καλλιέργεια. Δεν θα είναι αυτό το αποφασιστική σημασία στοιχείο δεν θα είναι αυτό που θα δώσει δυνατότητα να κάνουν, να λάβουν κάποιες πρωτοβουλίες σημαντικές. Γι' αυτό υπάρχει συνένεση τώρα σε σχέση με την αλλαγή του συστήματος για το όπως ισχύει σήμερα. Αν κάνει όμως ο καθένας ό,τι επιθυμεί, στο τέλος τέλος θα έχουμε τον κίνδυνο σε κάθε κράτος μέρος να έχουμε διαφορετικό σύστημα. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια κοινή αγροτική πολιτική πανευρωπαϊκά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόρφμαν ε, για τη ε, δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό. Θα μπορούσα να στηρίξω οτιδήποτε απλουστεύει τα πράγματα ε και μειώνει το διοικητικό άχθος. Αυτό είναι σημείο κίνησης. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εθνικό φάκελος για τις χώρες και εντός του φακέλου αυτού μπορούν να αποφασίσουν ε, πώς ε, θα ρυθμίσουν τις πληρωμές. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι προτάσεις του κυρίου Ντόρφμαν τροποποιούν το συνολικό φάκελο που είναι διαθέσιμο στις χώρες, αλλά εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής των εθνικών τους προγραμμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλή ε, διασύνδεση ανάμεσα ε, στις ε, εθνικές ας πούμε, προοπτικές και τις άλλες. Δηλαδή μπορεί στο Single Payment Scheme να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι πρόβλημα και για τις ε, υπηρεσίες που κάνουν τις πληρωμές. Κατανοώ βεβαίως ε, τις ανησυχίες ε, που έχουν οι χώρες για την ημερομηνία της 1ης Δεκεμβρίου και νομίζω ότι ο κύριος Ντόρφμαν επέτυχε εδώ μια καλή συμφωνία. Ένα καλό συμβιβασμό και τον συγχαίρω γι' αυτό τέλεια, αν μπορούμε να βρούμε κάτι που να το στηρίξουμε όλοι, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Τελικό σημείο. Σημείωσα ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για την χρηματοδότηση κτλ. Ο κύριος Ντόρφμαν έβαλε έτσι μία περίεργη φρασούλα ε, στην, επεξηγηματική του έκθεση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σχετικό, δηλαδή γίνεται αναφορά στην εκρίζωση και τα, και τα θέματα ε, πρόθεσης της καλλιέργειας. Ε, δεν νομίζω ότι έχει σχέση Πολλοί μεταξύ ημών πιστεύουν ότι ε, θα πρέπει να καταργηθούν ε, τα καλλιεργητικά δικαιώματα ε, και επομένως εδώ θα πρέπει να το συζητήσουμε πριν αποφασίσουμε να το βάλουμε στην έκθεση. Κυρία Κλάς, ναι, πρόεδρε, πραγματικά μεγάλους επένους προς τον Herbert Dorfman που το περίπλοκο θέμα προσπαθεί να το δαμάσει στην έκθεσή του. Και έτσι κατάλαβα και εγώ και τον συνάδελφο Καπόλα Σάντας. Γιατί να βιαστούμε με τέτοιες αποφάσεις. Στο συνολικό πακέτο με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2012 θέλει να αποφασιστούν όλα αυτά εφέτος υποχρεωτικά όταν τα άλλα θέματα εκκρεμούν για την ΚΑΠ ακόμα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά κάτι στους συναδέλφους ότι έχουμε και την κοινή οργάνωση αγοράς για τον ίνο και ιδιαίτερα με τέτοιο τρόπο τον έχουμε όπως το αποφασίσαμε με πολλούς, πολλούς κόπους καταφέραμε στην Ευρωβουλή να συμφωνήσουμε και να λειτουργεί έτσι και θεμελιώνεται και βασίζεται ότι στην μεταρρύθμιση της αγοράς για τον Ίνο δημιουργήσαμε αυτούς τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τα εθνικά χαρτοφυλάκια για τον Ίνο. Εθνικά τα κράτη-μέλη μπορούν ξεχωριστά να αποφασίζουν αν θα ενεργοποιηθούν και αν θα δράσουν για την ινοποιητική δραστηριότητα ξεχωριστά. Αυτό διαφοροποιεί τα πράγματα σε σχέση με την ΚΑΠ. Τώρα όμως σε μια απογραφειοκρατικοποίηση τι γίνεται, εντάσσεται η ινοποίηση σε αυτό το μεγάλο πακέτο των μέτρων μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Το πετάνε δηλαδή μέσα σε ένα καζάνι και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα από αυτή την ισοπαίδωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει, αλλά τίθεται το ερώτημα το οποίο αναφύεται και θα πρέπει να απαντηθεί όπως και αναφέρθηκε και πιο πριν. Όπως ε, αγαπητοί Χόισλινγκ είναι απόλυτα σημαντικό και για τους συνοποιούς αμπελουργούς της χώρας μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το χαρτοφυλάκιο, αυτός ο προϋπολογισμός, η ΚΟΑ, Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον Ίνο να παραμείνει ως έχει. Θέλουμε και στο μέλλον να είμαστε καινοτόμοι και με κάποιο εφάνταστο τρόπο να δημιουργήσουμε κάτι για την Ινοποία. Αυτό το πλαίσιο είναι η ΚΟΑ για τον Ίνο. Και από ό,τι βλέπω, η πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέρα από αυτό ανοίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα τη δυνατότητα η να εντάσσεται στο πριμ, στο συνολικό πριμ για, την, για τις καλλιέργειες, για την έκταση των καλλιεργειών. Σωστά το κατάλαβα, έτσι δεν είναι. Και ο συνάδελφος Ντόρφμαν τι θέλει. Θέλει εδώ να υπάρχει μια δυνατότητα τα κράτη-μέλη τα ίδια να μπορούν να αποφασίσουν αν θα εντάσσονται σε αυτό το σύστημα ή όχι. Εντάξει, αν είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα, αν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η πορεία Πρώτον, να πούμε δεν θέλουμε να ληφθεί απόφαση τώρα, προδικάζοντας τα πράγματα. Θέλουμε να αναμείνουμε, να αποφασιστούν οι υπόλοιπες προτάσεις για την μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής, να έχει ολοκληρωθεί και να έχει διευθετηθεί, να έχει αποφασιστεί έτσι για τις άλλες πτυχές και μετά θα αποφασίσουμε και για τον Ίνο και θα αφήσουμε τα θέματα στην εθνική αρμοδιότητα, δηλαδή ως θέμα των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ό,τι υπάρχει για την κοινή οργάνωση αγοράς ίνου θα παραμείνει άθικτο και θα παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν για τον προϋπολογισμό και τα κονδύλια για αυτή την κόα ίνου τα ίδια. Αυτά είναι τα τρία σημεία ως παρατηρήσεις που θα ήθελα να θέσω. Αν συμβαίνουν όλα αυτά τότε, πολύ σωστά τα διατύπωσε ο Herbert Dorfman στην έκθεσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κλάς. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον Χέρμπερ Τόρτμαν, να δώσω το λόγο στον Διευθυντή, τον κύριο Πατσέκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση. Πολύ σύντομα μπορώ να πω ότι δεν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με την έκθεση παρά μονάχα μία, μόνο που είναι σημαντική. Πριν από αυτό όμως ε, θα ήθελα να το αιτιολογήσω. Ε, το γιατί δηλαδή στην αρχική μας ε, πρόταση είχαμε προτείνει, είχαμε προβλέψει μονάχα μία ημερομηνία για την εθελοντική μετάβαση από την στήριξη που δίνεται ε, στον καλλιεργητή στην άμεση πληρωμή, στο σύστημα άμεσων πληρωμών. Είπαμε ότι καλύτερα θα ήταν να γίνει το 2012 έτσι ώστε να έχουμε το χρόνο να ετοιμάσουμε τα πάντα έτσι ώστε να μπορούν τις άμεσες πληρωμές να τις δέχονται μετά απευθείας οι γεωργοί. Εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι η ημερομηνία του Αυγούστου ως τελική ημερομηνία μπορεί να γίνει αποδεκτή. Να αποσαφηνίσω επίσης ότι ορισμένε χώρες μέλη έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την δυνατότητα μεταφοράς ε, των πόρων που διαθέτουν ε, στον αμπελοϊνικό τομέα προς τις άμεσες πληρωμές στο Λουξεμβούργο, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο το έχουν κάνει εξ ολοκλήρου, η Ισπανία και η Ελλάδα εν μέρη. Άρα βρισκόμαστε σε μεταβατικό κανονισμό και θέλουμε στο μεταβατικό υπογραμμίσιο κανονισμό να παραμείνει η κατάσταση ως έχει. Λοιπόν, θα σας πω τώρα την ε, δυσκολία που έχουμε και θα απαντήσω και στον κύριο Καπούλο Σάντος με την ευκαιρία. Δυσκολευόμαστε λοιπόν με την τροπολογία η οποία προδικάζει το τι θα ακολουθήσει το 2014 αυτό είναι ανοιχτό στην ε, συζήτηση. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις άμεσες πληρωμές και με την ε, μεταρρύθμιση της ΚΟΑ. Κατά την άποψή μου δεν με έχει θέσει μια τέτοια θεώρηση στον μεταβατικό κανονισμό. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην τροπολογία υπαριθμών 7. Κατά τα λοιπά κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα και επομένως μπορούμε εν τέλει να συμφωνήσουμε με την έκθεση και με όλα τα υπόλοιπα σημεία τα οποία σε αυτήν αναφέρονται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Ο Χέρμπερτ για να κλείσει η συζήτηση. Μάλιστα μια ολόκληρη σειρά ερωτημάτων και θεμάτων που θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω. Συμβαίνει όπως ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μόλις να έφερε. Δηλαδή, <clears throat> η σήμερα ενισχύει ρύθμιση για την αγορά ίνου προβλέπει ότι το εθνικό χαρτοφυλάκιο, ο εθνικός προϋπολογισμός εντάσσεται, μπορεί να περάσει στο σύστημα άμεσων πληρωμών. Και αυτό το έχουν κάνει κάποια κράτη-μέλη. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη ερώτηση της συναδέφου Λούλινγκ. Έτσι έχει γίνει αυτό. Όχι όμως έτσι όπως σχεδιάζουμε να γίνει στο μέλλον. Δηλαδή η προσωρινή αυτή τη στιγμή ένταξη έτσι, κάλυψη έτσι, σημαίνει ότι τα κονδύλια που υπάρχουν στο εθνικό χαρτοφυλάκιο στον προϋπολογισμό ανάγονται στην έκταση αμπελοκαλλιέργειας στα κράτη-μέλη άσχετα και ανεξάρτητα από τις ε, υπόλοιπες άμεσες πληρωμές. Αυτό οδηγεί για παράδειγμα στο ότι π.χ. για το Λουξεμβούργο οι άμεσες πληρωμές ε, για την αμπελουργία είναι πολύ ψηλότερες από ότι οι πληρωμές σε άλλους τομείς. Αυτό το σύστημα όταν σύστημα με, σύμφωνα με τις σημερινές προτάσεις ε, για την γεωργική πολιτική στο μέλλον δεν θα είναι εφικτό να λειτουργήσει έτσι. Θα υπάρχει είτε ένα εθνικό χαρτοφυλάκιο, δηλαδή εθνικός προϋπολογισμός, ή όχι ή, αλλά εν πάση περιπτώσει υποχρεωτικά η αμπελουργία θα εντάσσεται η εινοποιία στο κανονικό χαρτοφυλάκιο, στο σύστημα των άμεσων πληρωμών. Τώρα για μένα είναι φυσικά σαφές ότι με αυτή την τροπολογία υπαριθμών 7 του Ντέρεκ που οπωσδήποτε θα πρέπει να συζητήσουμε θα πρέπει να λάβουμε διαφοροποιημένα υπόψη συνολικό, στο συνολικό πακέτο να θέσουμε το ερώτημα και να δούμε τι θα κάνουμε. Πού, σε ποιο σημείο, πιο λογικά και με τον καλύτερο τρόπο μπορεί να ενταχθεί και να σχεδιαστεί. Είναι λογικό για όλους τους τομείς όλων των ε, εκτάσεων που καλλιεργούνται από πλευράς γεωργίας να γίνεται όταν υπάρχει μια κοινή οργάνωση αγοράς ε, με ίδια κονδύλια όπως για την εινοποιία θα πρέπει έτσι να εντάσσονται σε αυτό το σύστημα άμεσων πληρωμών ή όχι. Θα πρέπει να διατυπώσουμε αυτό το ερώτημα για να βρούμε την απάντηση. Και θα πρέπει να δούμε σε ποιο σημείο, με τον πιο λογικό και ε, πιο αποτελεσματικό τρόπο μπορεί να εξεταστεί μια τέτοια δυνατότητα πιο αποτελεσματικά. Αυτό ως προϋπόθεση, ως όρος. Και αυτό προϋποθέτει ακριβώς ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες ερωτήσεις αυτό προηγούμενο, με την ερώτηση της κυρίας ε, Ισπανίδα συναδέλφου απάντησα νομίζω με αυτόν τον τρόπο για την ερώτηση την παρέμβαση της κυρίας Άστριτ Λούλινγκ εν μέρη έχει απαντηθεί και στο σημερινό σύστημα το Λουξεμβούργο σήμερα ήδη ή και η Ισπανία δεν θα μπορούν στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο να λειτουργήσουν. Θα πρέπει να αποφασίσουν και να δούμε πώς άμεσα το σύστημα άμεσων πληρωμών θα λειτουργεί για την εινοποιία και πώς θα χρηματοδοτείται με κονδύλια από αυτόν τον προϋπολογισμό, τον ξεχωριστό προϋπολογισμό των κρατών μελών του Εθνικού Χαρτοφυλακίου ή με άλλα μέσα που θα διαθέτει ένα κράτος μέλος. Ναι, μετά στη συνέχεια ένα λεπτό. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που από πλευρά Χόισλινγκ αναφέρθηκε και από την συνάδελφο Κλάς προτάθηκε. Πιστεύω τα περισσότερα κράτη-μέλη με τα εθνικά χαρτοφυλάκια όσα έχουν σήμερα είναι ουσιαστικά πολύ ικανοποιημένα και δεν έχουν καμιά όρεξη, ας το πω έτσι, δεν θα ήθελαν η εινοποιία στο σύστημα άμεσων πληρωμών να ε, ενταχθεί με αρνητικές επιπτώσεις ή να υπάρξουν αλλαγές που δεν θα ήταν ευπρόσδεκτες και για τη συνολική συζήτηση αν θέλουμε ή όχι η νοποιία να εντάσσεται σε ένα σύστημα άμεσων πληρωμών ή όχι και για το θέμα των δικαιωμάτων φύτευσης ή εμφύτευσης και πάλι σε συνεννόηση με τον ε, εισηγητή μας ε, τον Μισελ Νταντάν απέφυγα στη δική μου έκθεση να κάνω λόγο και να τοποθετηθώ για τα εμφυτευτικά δικαιώματα και σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν που όμως δεν βρίσκεται σε αυτό το κείμενο αλλά σε συνοδευτική έκθεση που αναφέρεται ότι το Κοινοβούλιο τοποθετείται υπέρ των εμφυτευτικών δικαιωμάτων. Αυτό αληθεύει επειδή στην έκθεση δεν το είχαμε έτσι. Και ο συνάδελφος ε, Μισελ θα θυμάται ότι έχοντας συζητήσει αυτό το θέμα μαζί του το εντάσσεται στη δική του έκθεση για την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου και για το αν θα υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ ή κατά των εμφυτευτικών δικαιωμάτων για την εινοποιία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τίθεται. Το θέμα της συναδέλφου Κλάς για τις αποφάσεις ε, είναι τεχνικό θέμα το αν θα μεταφερθεί ή θα διατίθενται κονδύλια έτσι όπως από το Λουξεμβούργο. Ένα ένα μέρος αυτών των δυνατοτήτων ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας πενταετούς περίοδου που θα εκπνεύσει ή εκπνέει. Και πρέπει έτσι λοιπόν για το 2013 ή το 2014 μέχρι τότε να έχουμε μια προσωρινή μεταβατική ρύθμιση είναι τεχνικού χαρακτήρα θέμα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε μια μεταβατική ρύθμιση ώστε από το 2014 ας το πω έτσι να μπορούμε να λειτουργήσουμε μέχρι τότε χωρίς να εκκρεμούν αυτά τα θέματα και να μένουν μετέωρα εν κενό. Μετά θα έλεγα και ολοκληρώνω με αυτό και θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά. Έχω την εντύπωση που αποκόμισα ότι όταν τα κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη δίνεται η δυνατότητα που τους παρέχεται ένα τμήμα, ένα μέρος του εθνικού χαρτοφυλακίου του εθνικού προϋπολογισμού να το χρησιμοποιούν για το Single Payments Act και ταυτόχρονα υποχρεούνται υποχρεωτικά πρέπει να ε, κάνουν χρήση του δικαιώματος πριν ε, για τις εκτάσεις η πίεση από τον υπόλοιπο τομέα για την γεωργία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη στο τέλος τέλος τι θα γίνει. Οι τελικές επιπτώσεις, όχι πρόθεσμα αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε πολλά κράτη-μέλη αυτό το εθνικό πλαίσιο χαρτοφυλακίου θα οδηγήσουν στο να εξαφανιστεί και να περάσουμε σε ένα σύστημα άμεσων πληρωμών. Θα έπρεπε πραγματικά να θέσουμε στον τομέα αυτό το ερώτημα. Έχει νόημα να γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Και υπό το πρίσμα του σημείου στην ημερήσια διάταξη όπω το είχαμε εντάξει. Εθνικό χαρτοφυλάκιο, εθνική προπολογισμή και με τα μέτρα και κονδύλια σε σχέση με αυτές τις δράσεις συνεισφέρει να είναι ένας ανταγωνιστικός τομέας ο τομέας της ευρωπαϊκής συνοποιίας στην Ευρώπη και παγκόσμια. Πρόκειται για το θέμα αυτής λοιπόν της αηφορίας της ε, ανταγωνιστικότητας, ε, της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας. Τι θα κάνουμε λοιπόν, δεν θα βοηθήσουμε στην, τον εινοποιητικό τομέα. Αν δίνουμε πριμ αναέκταση για την εινοποιία για την αμπελουργία, αλλά όμως ε, δεν υποστηρίξουμε με εθνικά ή ειδικά μέτρα την εινοποιία και καταργηθεί το εθνικό πλαίσιο, ε, το εθνικό χαρτοφυλάκιο. Πρέπει λοιπόν, μια και είναι ένας από τους πιο ενεργούς τομείς της γεωργίας, σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουμε υπόψη αυτό. Δεν εξυπηρετούμε καθόλου εξαφανίζοντας αυτά τα κονδύλια των εθνικών χαρτοφυλακίων και των ειδικών μέτρων τα κράτη-μέλη για την εινοποιία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούλινγκ θέλει μια σύντομη απάντηση. Μία ακόμη ερώτηση, αν κατάλαβα καλά εάν ο εθνικός φάκελος ενσωματωθεί στο Single Payment Scheme τότε θα επηρεαστεί από το flattening, δηλαδή από την εξομοίωση, την ισοπαίδωση. Ο εθνικός φάκελος που ενσωματώνουμε θα αυξήσει τον προϋπολογισμό στον πρώτο πυλώνα, τουλάχιστον στις συνοπαραγωγούς χώρες. Και θα πρέπει να εξισορροπήσουν ακόμη περισσότερο, δηλαδή να μεταφέρουμε ακόμη περισσότερο προς τα κράτη-μέλη, τα οποία λαμβάνουν λιγότερο. Δηλαδή, η αμπελουργία θα χάσει μέγα μέρος του χρηματοδοτικού της φακέλου. Αυτό δεν είναι φαντασιοπληξία, είναι πραγματικότητα. Με αριθμούς ε, κατανοούμε και συνενούμαστε καλύτερα. Και έχουμε και αριθμούς ε, σε σχέση με το κράτος Το εθνικό χαρτοφυλάκιο ήταν περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ ετήσια. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό και για μέτρα του Εθνικού Χαρτοφυλακίου όπως έχουν αποφασιστεί για την κοινή οργάνωση αγοράς χρησιμοποιούνται. Και αν θέλει ένα κράτος μέλος μπορεί αυτό να ισχύει και στο μέλλον. Έτσι να εφαρμόζεται. Ταυτόχρονα όμως αποφασίζουμε και εγκρίνουμε στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ότι η εινοποιία θα είναι επιδοτήσιμη καλλιέργεια. Αν υποθέσουμε ότι το μέσο ποσό θα είναι περίπου για την Ιταλία 300 ευρώ επί 600.000 εκτάρια εινοποιίας 180 εκατομμύρια ευρώ. Τίθεται το ενδιαφέρον ερώτημα και το κατανοώ βέβαια υπό το πρίσμα των εινοποιών και εγώ θα το έλεγα ότι θα επιθυμούσα το εθνικό χαρτοφυλάκιο να διατηρηθεί με τα 220 τόσα και μετά να καταβάλλονται και τα 180 εκατομμύρια. Όμως ο κανονισμός αυτός δεν το αποκλείει αυτό ως δυνατότητα. Όμως αυτά τα 180 εκατομμύρια του πρώτου πυλώνα από κάπου πρέπει να προέλθουν. Δεν είναι έτσι διαθέσιμα χίδιν, προέρχονται από άλλους τομείς της γεωργίας. Και γι' αυτό λέει αυτός ο, η κλωνοποίηση. Μπορείτε κράτη-μέλη να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέρος του εθνικού προϋπολογισμού στο εθνικό χαρτοφυλάκιο. Ώστε αυτά τα κονδύλια αυτές οι άμεσες πληρωμές να εντάσσονται για τη χρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα. Μπορεί το κράτος μέλος να λάβει αυτή την απόφαση. Τα 180 εκατομμύρια του Εθνικού Χαρτοφυλακίου έτσι να τα πάρει και να τα περάσει στο σύστημα άμεσων πληρωμών. Δεν θα το κάνουν όμως, δεν θελήσουν να το κάνουν οι νοποιοί. Οι υπόλοιποι γεωργοί θα θελήσουν να το κάνουν. Διότι για αυτά τα 180 εκατομμύρια ευρώ που λείπουν από τους άλλους γεωργούς. Και γι' αυτό για τα πριμ στον πρώτο πυλώνα το πριμ είναι χαμηλό, είναι μικρό. Αλλά αν γίνει αυτό θα υπάρξει μεγάλη πίεση στον τομέα της συνοποίησης του εθνικού, για το εθνικό χαρτοφυλάκιο. Να χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια στο σύστημα άμεσων πληρωμών. Εκεί να εντάσσονται. Και αυτό θα σημαίνει το τερματισμό, το τέρμα, την εκπνοή των εθνικών χαρτοφυλακίων και εθνικών προπολογισμών. Και αυτό δεν το θεωρώ σκόπιμο για τον εινοποιητικό τομέα και γιατί θα έπρεπε για την εινοποιία να την εντάξουμε υποχρεωτικά στον πρώτο πυλώνα και να έχουμε την πριμ, πριμοδότηση όσον αφορά την έκταση, την καλλιεργούμενη έκταση υπό τον πρώτο πυλώνα. Αυτά είναι τα επιχειρήματα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε όλες μας τις αμφιβολίες. 1η Ιουνίου στις 12 τροπολογίες. Αν δεν έχετε άλλες τοποθετήσεις, πάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο. Πω ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και πρόθεσή τους, μια στρατηγική για την πρόθεση των γεύσεων της Ευρώπης. Θα ακούσουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν ε, για την στρατηγική, για την πρόθεση των γεύσεων της Ευρώπης. Η έκθεση είναι του Ζωζέ Μποβέ και του δίνω το λόγο. Ζωζέ, έχεις το λόγο. μέτρα πρόθεσης για τα προϊόντα ποιότητας, ποια στρατηγική για την πρόθεση των γεύσεων. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, είδε, γεννήθηκε αυτή η έκθεση ε, είναι, το, είναι η πράσινη βίβλος της Κομισιόν και η ανακοίνωση του Μαρτίου 2000 12 για την πρόθεση των γεύσεων. Όλα αυτά πρέπει να καταλήξουν σε το, τον, το φθινόπωρο του 2012 σε μία πρόταση. Τώρα, πού τοποθετούμεθα και γιατί συζητάμε και από πού ερχόμαστε. Από μία πρώτη πολιτική της δεκαετίας του 80, όπου η πρόθεση των προϊόντων γινόταν μόνο και μόνο για να καταναλωθεί το πλεόνασμα. Δεν ήταν δηλαδή ένα θέμα ποιότητας, αλλά ένα θέμα αποσυμφόρησης των αγορών. Διαχείριση των πλεονασμάτων λοιπόν. Το 2000 είχαμε μία εξέλιξη αυτής της πολιτικής, διότι υπήρξε και ένα σχετικός έλεγχος των, ε, των της παραγωγής δεν είχαμε δηλαδή αντίστοιχες καταστάσεις, αλλά μετά είχαμε αυτά τα γνωστά σκάνδαλα, ε, διοξίνη στα αυγά, τρελές αγελάδες. Πέρυσι θυμηθείτε τα, ε, τα, Και όλα αυτά τα θέματα λοιπόν έχουν, ε, ε, οι έχουν ως στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τον καταναλωτή για να μπορέσει να αρχίσει να καταναλώνει τα προϊόντα τα οποία είχαν πληγεί από τα σκάνδαλα. Αυτή ήταν η παλιά πολιτική του 2000. Τώρα, όταν διαβάζουμε εμείς αυτά τα οποία μας λέει η Κομισιόν, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια νέα πια λογική. Διότι στόχος είναι να εφαρμόσουμε στρατηγικές για να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία στην τροφιμική αλυσίδα χρησιμοποιώντας την πρόθεση και την πληροφόρηση μέσα στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής. Έχουμε λοιπόν τέσσερα θέματα τα οποία προτείνονται από την Κομισιόν πραγματική προστιθέμενη αξία και δημιουργία αυτή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, βελτίωσης των προγραμμάτων πρόθεσης, αποτελεσματικότερα ε, προγράμματα και συνέργεια μεταξύ των διαφόρων μέσων πρόθεσης που έχουμε. Αυτές είναι οι γενικές θεματικές που προθούνται. Ο προϋπολογισμός παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα ταπεινός. Έχουμε 55 εκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον στόχο. Χρειάζεται μία συγχρηματοδότηση σήμερα. Είναι ένα σύστημα αρκετά πολύπλοκο και έχουμε έναν προϋπολογισμό αρκετά μειωμένο. Το 70% αυτού του προϋπολογισμού καταναλώνεται μέσα στην Ευρώπη και έχει ως στόχο την επέκταση αυτής της πρόθεσης προς ε, τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού βρισκόμαστε σήμερα και προς τα πού πρέπει να τίνουμε. Αυτός είναι ο στόχος της έκθεσής μου. Εμείς ε, θεωρούμε σε επίπεδο έκθεσης ότι οι προτάσεις της Κομισιόν πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά θα έπρεπε όμως να προχωρήσουμε και πιο, πιο μακριά. Δηλαδή, για τον ορισμό της ποιότητας και της ποικιλότητα ε, των, των ευρωπαϊκών ε, τροφίμων. Διότι στην πρόταση της Κομισιόν μιλάμε για γεύσεις της Ευρώπης εμείς δεν ξέρουμε τι θέλει να πει καλά-καλά αυτός ο όρος. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτήν, αυτόν τον πλούτο, την διαφορετικότητα, την ποικιλία των γεύσεων και προελεύσεων των προϊόντων. Αυτές είναι οι βασικές έννοιες για να ξέρουμε περί τίνος μιλάμε. Δηλαδή γεύσεις της Ευρώπης, στον πληθυντικό και όχι στον ελληνικό. Σήμερα έχουμε μερικά συγκεκριμένα στοιχεία για την ποιότητα που μπορούν να αποτελέσουν βάσεις. Είναι οι ειδικές, ε, τα ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται από την προέλευση, την παράδοση, τα πολιτιστικά και τον τρόπο παρασκευής. Ε, έχουμε τις ε, γεωγραφικές προελεύσεις, παραδοσιακές και σε εγγυημένες παραγωγές και πρέπει να ξεκινήσουμε από, αυτού, από αυτήν την αρχή του, από αυτόν τον πρώτο ορισμό να καταλήξουμε σε αυτές τις περιφερειακές γεύσεις που ορίζουν τη διαφορά των γεύσεων και όχι στις μεγάλες μάρκες που έχουν ομοιογενοποιημένες γεύσεις. Τώρα, πέρα από αυτή την πολιτική γεύσεων και ορισμών τους ε, και όσον αφορά το τερουάρ και τις πρακτικές, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ε, μία καλύτερη ανταμοιβή ε, των παραγωγών, δηλαδή όλη αυτή η ποιότητα κάπου θα πρέπει να ανταμείβει τους γεωργούς. Πρέπει να προχωρήσουμε βέβαια πέρα και πέρα από αυτό. Αυτό πρόκειται για την αφετηρία. Εγώ στην έκθεσή μου θα προεπιστώ την ιδέα να προωθήσουμε πέρα από αυτά τα πρώτα στοιχεία και τα διάφορα συστήματα αηφορίας στην παραγωγή που να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις των γεωργών, διατήρηση και υπεράσπιση της βιοποικιλότητας, πολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει δηλαδή να εντάξουμε νέα στοιχεία όπου βλέπουμε ότι τελικά οι Ευρωπαίοι Γεωργοί ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και θα ήμασταν έτσι και σύμβατοι με τα προγράμματα τα οποία ξεκίνησε η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα δεν πρέπει κανείς να έχει την αυταπάτη ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής. Αυτό δεν έχει νόημα. Έχουμε μια διαφορετικότητα στη γεωργία. Δεν μπορούμε να τα μπερδεύουμε όλα αυτά και να λέμε υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, διότι σήμερα αυτό θα εξαπατούσε τον καταναλωτή. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σαφείς και να έχουμε μία πιο σαφή αντίληψη. λέμε ότι τίνουμε προς μία πιο απλή διαχείριση, μία συνέργεια στα προγράμματα, αυτό είναι, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί ως προς τους όρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέταρτο σημείο της ανακοίνωσής της λέει κάτι το οποίο είναι σημαντικό και τονίζει ένα σημείο που για μας είναι απόλυτα συνεκτικό με τα άλλα σημεία τα οποία υπογραμμίσαμε και το αναφέρω, σημασία των τοπικών αγορών, η, η σύντομη μικρή ε, τροφιμική αλυσίδα, η ευημερία των ζώων, οι φόροι, τρόποι παραγωγής και άλλα. Πρόκειται λοιπόν για ε, σημαντικά στοιχεία τα οποία λειτουργούν προσθετικά σε όλα όσα σας έλεγα πριν. Και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ευρωπαϊκού μοντέλου παραγωγής. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο μεταξύ των τοπικών παραγωγών και με αυτές τις νέες προκλήσεις και να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Αυτή είναι η διομορφία. Σε αυτό θα βασιστεί η δουλειά μου. Η αποδοχή ε, στα προγράμματα θα περνάει από το σεβασμό αυτών των στοιχείων και μετά θα πρέπει να είμαστε και συνεπείς ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και στις τρίτες χώρες, ε, να στείλουμε μάλλον και στις τρίτες χώρες ένα μήνυμα για να μπορέσουν να καταλάβουν πώς αυτά τα προϊόντα ανταποκρίνονται σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Αυτά είναι τα διάφορα σημεία τα οποία θα αναπτύξω. Θεωρώ ότι αυτό το μέσο θα πρέπει να καταστεί ένα ευρωπαϊκό μέσο για την ευρωπαϊκή παραγωγή και τις ευρωπαϊκές γεύσεις, να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ γεωργίας και της παραγωγής και των καταναλωτών. Διότι αυτό θα επιτρέψει στους γεωργούς να έχουν και ένα καλύτερο εγγυημένο εισόδημα και οι καταναλωτές να έχουν και αυτοί μια δίκαιη τιμή για το προϊόν που αγοράζουν. Πρόκειται για κάτι το οποίο τίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, θα προτείνουμε όμως και άλλες βελτιώσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ο Κοσμάκης να μας καταλαβαίνει και να βγαίνουμε και από αυτή την αμφισημία των διαφόρων πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ. Ζωζέ, ξεκινάμε τη συζήτηση. Ε, Ράνς Καρσία και μετά κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ καλή η δουλειά του κυρίου Μποβέ, διότι είναι κατεπίγουσα η πρόταση της Κομισιόν. Είναι απαραίτητη για την κοινοτική παραγωγή, αλλά και για τους καταναλωτές. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αγνοούν την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παραγωγής. Δεν καταβάλαμε ποτέ την προσπάθεια για να εξηγήσουμε τις ονομασίες προέλευσης, τις, τα παραδοσιακά προϊόντα, τη γεωγραφική προέλευση, δεν την εξηγήσαμε στον καταναλωτή. Είναι πολύ απαραίτητο κάτι τέτοιο. Για την προστιθέμενη αξία της, ε, ό,τι είναι υπέρ της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής παραγωγής είναι πρόσδεκτο. Σε αυτά τα κεφάλαια της ε, Κομισιόν για, τα γενικά προ... για την ε, περίπτωση κρίσης και την πρόθεση των προϊόντων σε περίπτωση κρίσης. Πριν από ένα χρόνο ξέσπασε το σκάνδαλο του Εκόλη που ξεσήκωσε τον κοινοτικό πληθυσμό απίστευτα. Αλλά κυρίως ήταν σκανδαλώδης και η επίθεση ε, κατά των κοινοτικών προϊόντων χωρίς να υπάρχει και κανένας λόγος. Πώς θέλει η Κομισιόν εμείς να την πιστεύουμε μετά από όλα αυτά που τραβήξαμε πρόσφατα. Ε, εγώ θα ήθελα ταχύτητα στη δράση. Δεν αξίζει δηλαδή μήνες μετά, ένα χρόνο, δύο χρόνια μετά να κάνουμε διαφήμιση της παραγωγής, διότι η ζημιά έχει γίνει πια και δεν δε, δε, δε, γλιτώνει. Πώς ε, θα πλουστεύσει τις διαδικασίες η Κομισιόν ούτως ώστε αυτό το χρήμα σε περίπτωση κρίσης να είναι χρήσιμο. Άλλο, <coughs> τα ζητούμενα για τους ενδιαφερόμενους για να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια. Πώς μπορεί να είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή κάθε φορά που η Κομισιόν προτείνει να, βγάζει, να αφαιρεί γραφειοκρατία ή να διευκολύνει τα πράγματα, τι διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα μπερδεύονται 10 φορές παραπάνω. Ποια είναι η ιδέα της Κομισιόν που σας δίνει, κύριε σας δίνει η Κομισιόν καμιά ιδέα κύριε Μποβέ ή εσείς μπορείτε να δώσετε καμιά ιδέα στην Κομισιόν. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, από ό,τι κατάλαβα θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα προώθησης. Εγώ ρωτώ με τι παράδες είναι το, θα είναι τα ίδια λεφτά με αυτά τα οποία, τα οποία έχουμε σήμερα ή θα βρει η Κομισιόν αλλού κονδύλια για να αντιμετωπίσει όλη αυτή την ε, διαφημιστική καμπάνια. Για το κρασί, που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται τρόφιμο, υπόκειται διακρίσεις έναντι των άλλων τομέων, διότι απαγορεύεται η πρόθεση του κρασιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κοινοτικά κονδύλια. Να είμαστε γενναίοι κύριε Μποβέ, σας προτείνω Ας κοιτάξουμε τουλάχιστον στις χώρες εκείνες όπου το κρασί θεωρείται τροφή, να επεκτείνουμε την πρόθεσή τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω αποκλειστικά στις χώρες εκείνες όπου το κρασί θεωρείται τροφή. Θα έχουμε ισότητα και δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ η κυρία Γιούζο και μετά Πετράου Νέβες. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Γιούζο. Gracias, presidente. Bueno, no, le decía que las adoro. Έλεγα ότι η σκιώδης η δεν μίλησε ακόμη και είναι η κυρία Πατράου και να πάρω εγώ το λόγο στη συνέχεια. Τι λέτε κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε. E Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευγένεια και ζητώ συγγνώμη για αυτή την σύγχυση και κυρίως με το μικρόφωνο αυτό που δυσχέρανε την κατάσταση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή είναι και το πρώτο σημείο το οποίο μέσα σε ένα νέο πλαίσιο που τίθεται το θέμα αυτό για μένα είναι θεμελιώδους σημασίας στο ιστορικό πλαίσιο που είχαμε αλλά σήμερα έχουμε ένα νέο καινοτόμο πλαίσιο το οποίο μας δείχνει ότι αυτή η πορεία είναι που πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή είναι η πορεία που συμφωνούμε επ' αυτής όλοι πέρα από κάποια εξειδικευμένα συγκεκριμένα θέματα που θα τεθούν και πρέπει να αποφασίσουμε και να ρυθμίσουμε αλλά εδώ τίθεται το θέμα των προϊόντων που πρέπει να εντάσσονται δηλαδή της γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ευρώπη, συμφωνούμε όλοι γι' αυτό. Αλλά είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ότι αυτή η νέα λογική, όπως λέει ο κύριος Μποβέ, να δούμε αν αυτή η πορεία θα ανταποκριθεί στο κυριότερο αίτημα. Αξίζει τον κόπο το θέμα το οποίο τι θέτουν οι γεωργοί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και για το οποίο θέμα δεν έχουμε ακόμα απάντηση. Αξίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τέτοια μέτρα μέτρα τα οποία θα είναι τόσο απαιτητικά και σκληρά όσον αφορά υγειονομικές προϋποθέσεις για την υγεία, περιβάλλον, ευζοία των ζώων, σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτά τα οποία θα επιβάλλονται για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους ώστε να μπορούν να έχουν και υψηλότερο κόστος παραγωγής αυτά τα προϊόντα από πλευράς μας. Αξίζει τον κόπο ή όχι να υπομισθούν όλους αυτούς τους κανόνες και να ε, συμμορφωθούν με αυτούς οι παραγωγή μας. Αν με αυτή την έκθεση καταφέρουμε να καταδείξουμε ότι είναι εφικτό να αυξήσουμε, να έχουμε πρόσθετη αξία για τα προϊόντα που παράγουν οι δικοί μας γεωργοί και κτηνοτρόφοι και στην εσωτερική αγορά αλλά και στην εξωτερική αγορά, ε μάλιστα κύριοι, για πρώτη πρώτη φορά θα έχουμε μια απάντηση που θα αξίζει τον κόπο αυτό το εγχείρημα. Αν όχι, αν δεν το καταφέρουμε θα παραμένει πάντα το ίδιο ερώτημα. Πώς θα κερδίσουμε τη μάχη, των αγώνα της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τα έξοδα τις τιμές προϊόντων που θα είναι αυξημένες. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα που πρέπει να θέσουμε. Είναι η μεγάλη ευκαιρία που έχουμε τώρα εδώ ενώπιόν μας να μπορέσουν τα προϊόντα των παραγωγών μας με όλους αυτούς τους κανονισμούς να καταφέρουμε να επιβιώσουν στην αγορά και να μπορέσουμε να είναι ανταγωνιστικά και να υπάρχει αντιστάθμισμα για το κόστος, για το πρόσθετο κόστος, για όλους αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς που θα πρέπει να υπομισθούν. Πέρα από όλα αυτά υπάρχουν εδώ κάποιες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω πέρα από τα όσα ανέφερα ότι συμφωνώ με αυτό το οποίο λέει ο εισηγητής και με αυτό το οποίο η συνάδελφος ε, η Εστέρ είπε πιο πριν ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν πράγματι de facto στην έκθεση αυτή που θα εκφράζει συνενετικά τις θέσεις της Επιτροπής μας για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν για τη συζήτηση να προσθέσω για τη συζήτηση κάποιες πτυχές που θεωρώ ότι είναι και αυτές σημαντικές. Πρώτον, η πρώτη πτυχή, να κατανοήσουμε απόλυτα σαφώς ότι αν εμείς εδώ και πολύ χρονικό διάστημα αγωνιζόμαστε για την ποιότητα και πολυμορφοποίηση των προϊόντων μας είναι μια μάχη που κερδίζουμε και πρέπει να κερδιθεί και γι' αυτό είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε μια καλή θέση στην αγορά για αυτά τα προϊόντα. Η μία πτυχή δεν θα αντισταθμίσει στην άλλη, το ένα δεν α, απαλήφει το άλλο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ανταγωνιστικότητα στο εξωτερικό να κερδίσουμε στις εξωτερικές αγορές τις αναδιόμενες αγορές των αναδυόμενων κρατών και στην Ευρώπη πρέπει να το δούμε αυτό θέλουμε καλύτερη κερδοφορία των προϊόντων μας μεγαλύτερες αγορές που θα είναι διαθέσιμες για αυτά τα προϊόντα τότε πρέπει κάτι να κάνουμε για να ανοίξουν αυτές οι αγορές και να υπάρξει η δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων μας σε μεγαλύτερη κλίμακα με τις αναδιόμενες χώρες και αγορές πώς θα είμαστε σε θέση να θέσουμε τα προϊόντα μας, προϊόντα μας σε αυτές τις νέες αγορές και πώς θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των επιχειρήσεών μας ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες αγορές με τα προϊόντα τους. Απλούστευση και εξαπλούστευση. Μιλήσαμε και γίνεται πολλή λόγος γι' αυτό. Πώς θα τα καταφέρουμε και ο προπολογισμό και όλα αυτά αναφέρθηκαν, όλα αυτά τα έχουμε στα χαρτιά μπροστά μα. Τι θα αλλάξει, τι θα αλλάξει αν δεν έχουμε πραγματικά έναν προϋπολογισμό υποστήριξης, ενισχυτικό προϋπολογισμό, για να πάρουν ε, διαμόρφωση πραγματικά και να λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα για τα οποία συζητούμε και συμφωνούμε επαρτούν σε αυτή την έκθεση. Χρειάζεται κάποια αύξηση των κονδυλίων που συνδέονται με αυτούς τους τομείς, γιατί διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Μια άλλη πτυχή που και εδώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και αυτή. Οι παραγωγοί μας χρειάζονται εκείνοι που θα είναι υποψήφοι για να ενταθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα χρειάζονται πραγματικά απλούστευση κανόνων πρόσβασης. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σαφή κριτήρια για την πρόσβασή τους προς πελασιμότητα σε αυτές τις διατάξεις και να είναι διευκολυμένη η προσπελασιμότητα. Για εκείνους που δεν θα το καταφέρουν δεν θα σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες και να διερευνήσουν δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων τους ε, για τις εξωτερικές, τις αγορές στο εξωτερικό και με μεγαλύτερη κερδοφορία. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι διάσημα, διαθέσιμα τα αναγκαία στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξαγωγές, πληροφορίες για επαφές, ε, για κομβικά σημεία, για εξαγωγές, ε, διεργασίες και διαδικασίες, ένα εγχειρίδιο, ένα βιβλιάριο το οποίο θα μπορούσε να συνταχθεί για να εξυπηρετεί τις ενώσεις παραγωγών, τους παραγωγούς, για να διευκολύνονται αυτές οι διεργασίες διάθεσης των προϊόντων τους, για να μπορέσουν πραγματικά να διαθέσουν και να στέλνουν τα προϊόντα τους σε μια μεγαλύτερη εξωτερική αγορά με πρόσθετη αξία και κέρδος και κερδοφορία. Επίσης το θέμα των προκαταβολών και αυξημένων προκαταβολών, μια και έχουμε μεγάλους όγκους χρηματοδοτικούς εδώ και το 30% του κόστους, του ετήσιου κόστους δεν επαρκεί πάντα ώστε να ξεκινήσουμε τέτοιου είδους μεγαλόπνοα και μεγάλα, μεγάλης κλίμακα σχέδια να δώσουμε κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν κατηγοριοποιήσεις, ομαδοποιήσεις να υπάρξει και μια συγκεκριμένη κριτική κρίσιμη μάζα για να μπορούμε να, να, έχουμε συναλλαγές με, την, με τις αγορές σε παγκόσμια κλίμακα και πιλωτικά προγράμματα σε σχέση με τρίτες χώρες για το άνοιγμα και εκμετάλλευση αγορών και γενικούς, σε γενικούς όρους πέρα από αυτά τα μέτρα και κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να εξετάσουμε δεν θέλω να, χρονο, μακρηγορήσω αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ώστε μέσα σε αυτή τη νέα λογική για την οποία κάνατε λόγο και εμείς πρέπει να βρούμε μια νέα λογική για τις απαντήσεις. Αυτή η νέα λογική για τις απαντήσεις δεν μπορεί να είναι η παλιά μέθοδος για την παρουσίαση ιδεών. Πρέπει να συνεχίσουμε με προγράμματα δράσης αποτελεσματικά που θα μπορούν να διασφαλίζουν ότι τα δικά μας προϊόντα θα κερδίζουν, θα αποκτούν αυτή την πρόσθετη αξία και θα αναβαθμίζονται για να διατίθενται στις αγορές, για τη διάθεσή τους στις απαιτητικέ αγορές και τη διάθεσή τους με κερδοφορία. Ή θα το καταφέρουμε με αυτή την ευκαιρία ή δεν θα το έχουμε καταφέρει σε σχέση με τις ευθύνες μας έναντι των γεωργών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πατράου Πώς. Χάουαρντ μετά. Ευχαριστώ τον εισηγητή της και ο εισηγήτρε σήμερα όλα όσα είπε η κυρία Πατράου. Και για το πώς ονομάζεται το πρόγραμμα γεύσης της Ευρώπης είναι ένα σήμα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Το σημαντικό είναι να έχουμε τα προϊόντα μας μέσα. Η γεωργία μας έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την ευηρία των ζώων, με τη βιοπικιλότητα, με τα κοινωνικά μέτρα. Υπάρχουν χιλιάδες διατάξεις. Έχουμε τα πιο ασφαλή γεωργικά προϊόντα του κόσμου. Τι συμβαίνει. Είναι πιο ακριβά στην παραγωγή. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε και μέσα και έξω. Και φυσικά στον Ευρωπαίο καταναλωτή. Για παράδειγμα τα αυγά. Θέλουμε 750 τετραγωνικά εκατοστά κλουβί για, για τις κότες. Ε, αυξήθηκε η τιμή των αυγών και τι κάνουμε εμείς. Ε, εισάγουμε αυγά από τη Βραζιλία και τις Ηνωμένε Πολιτείες που, που τα κλουβιά είναι 350 τετραγωνικά εκατοστά. Μα τι μας νοιάζει εμάς αν οι κότες μας είναι οι πιο ευημερούσες κότες στον, ανά τον κόσμο όταν κανένας δεν το ξέρει. Εγώ συνεργάζομαι για να ζουν οι κότες όσο το δυνατόν καλύτερα. Το παλεύω. Αλλά πρέπει κανείς να το ξέρει. Υπάρχει μια έκθεση της ΕΦΣΑ στις 4 Απριλίου που λέει ότι αφού αναλύθηκαν πάρα πολλά προϊόντα, όλα τα εισαγόμενα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ε, ζυζανιοκτώνων έχουμε ένα σωρό κλάδους που τους παρατήσαμε από την καλλιέργεια διότι δεν μπορούμε να τους καλλιεργήσουμε άμα δεν τους ραντίσουμε. Και τα ίδια προϊόντα εμείς τα εισάγουμε από άλλες χώρες οι οποίες ραντίζουν. Εμένα πολύ ωραία όλα αυτά που λέει η Κομισιόν και το χρήμα βέβαια είναι λίγο, αλλά Πρέπει εμείς να κάνουμε εσωτερικές καμπάνιες πρόθεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξηγούμε γιατί τα προϊόντα μας είναι ακριβότερα και είναι καλύτερα. Και να ζητήσουμε να συνεργαστεί και ο ιδιωτικός τομέας και να υπάρχει διαφάνεια και όσο το δυνατόν πιο απλοί κανόνες. <coughs> Αλλά πρέπει να έχουμε τη συνέστηση ότι η γεωργία μας είναι πολύ πιο ακριβή από ό,τι αλλού. Άντε και για τις κονσέρβες, μην αρχίσουμε να μιλάμε για τις κονσέρβες ψαριών που έρχονται από την Νοτιοανατολική Ασία. Διότι δεν έχουν καν έλεγχο. Λοιπόν, αν δεν απαγορεύουμε εμείς την εισαγωγή αυτών των κονσερβών, να εξηγήσουμε τουλάχιστον γιατί τα δικά μα τα προϊόντα είναι καλύτερα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τώρα όσοι, όσα είπε και η κυρία Ράν για το κρασί, φυσικά είναι τρόφιμο το κρασί, είναι τροφή. Έχουμε ένα σωρό θέσει εργασία και στο μεταπητικό τομέα και στον πρωτογενή τομέα και πρέπει να συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ. Ωραία. Χόλουερτ και μετά Ντόρφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παίζει κεντρικό ρόλο η γεωργία στην οικονομία πολλών ε, χωρών μελών ε, και βεβαίως οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει την ε, ε, αύξηση των εξαγωγών, την αναγνωρισιμότητα, τη μεταπητική βιομηχανία που σχετίζεται με τα γεωργικά προϊόντα μας βρίσκει σύμφωνος. Στην χώρα μου ο τομέας της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων είναι ο πιο σημαντικός εγχώριος τομέας παραγωγής. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα νέα εμπορικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν λαμβάνοντας υπόψη και την παγκόσμια συγκυρία αυτή τη στιγμή ε, ε, ξαναβλέπουμε την ίδια ιστορία. Η ίδια η Κομισιόν έχει πει ότι, έχει αναγνωρίσει μάλλον ότι υπάρχει υπερβολικά μεγάλη γραφειοκρατία στην ε, Γεωργία. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς το έχουμε επανειλημμένα πει και στη δικιά μας Επιτροπή εδώ. Επομένως, οτιδήποτε είναι απλό και συνεκτικό και μπορεί να δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα και να μην παραμείνει μονάχα ευχές και ευχολόγια και λόγια, μας βρίσκει σύμφωνους θα πρέπει να απλουστευτεί η διαχείριση των ε, προγραμμάτων ε, εμπορίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο εισηγητής θέλει να προωθηθούν τα ε, ε, προϊόντα ποιότητας, αυτά τα οποία είναι ας πούμε λεγμένης προέλευσης, με ονομασία προέλευσης κτλ. Βεβαίως αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ε, οτιδήποτε αφορά τη μικρή γεωργία και την οικογενειακή εκμετάλλευση θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερα προς το προσοχής. Ε, προστιθέμενη αξία στην ΚΑΠ θα δώσει βεβαίως σε μια τέτοια αντιμετώπιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η γεύση της Ευρώπης να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την κατανάλωση ευρωπαϊκών προϊόντων. Γιατί εκεί ακριβώς και σε αυτή την παραγωγή κρύβονται πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Θα πρέπει να πρεθούν και διαδικασίες, διαργασίες οι οποίες σχετίζονται με την τοπική αγορά να καλυφθούν οι προσπάθειες αυτές από προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Ε, νομίζω ότι είναι αντιπαραγωγικό ε, να ξεκινήσουμε έτσι σε πολύ υψηλό επίπεδο κάποιες ε, εκστρατείες. Θα πρέπει να στοχεύσουμε αγορές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε one size fits all. Αυτού του είδους η πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον καθένα θα πρέπει να προωθήσουμε βεβαίως ε, σε εθνικό, ε, συγγνώμη, σε τοπικό επίπεδο την ανάπτυξη των προϊόντων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορούν τα τοπικά προϊόντα να συμμετέχουν στο εθνικό ε, πρόγραμμα ανάπτυξης. μικρο, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις σε πολλές περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες ε, παράγουν τέτοια ποιοτικά προϊόντα και θα πρέπει να στηριχτούν μέτρα προώθησης αποτελεσματικά όμως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία, εάν και εφόσον εφαρμοστεί σωστά, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην εξαγωγική προσπάθεια που κάνουν οι γεωργοί. Θα πρέπει πάντως να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα των δημόσιων προμηθειών ε, σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τέλος, ε, έχουμε συναντήσει τους εκπροσώπους ε, της ε, ε, και πρέπει να το ξανακάνουμε, να συναντήσουμε δηλαδή τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, γιατί θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες αυτό. Κατά τα λοιπά, ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ έγκαιρη και σωστή έκθεση. Herbert Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δύο ερωτήσεις. Ήδη μας είπε ο εισηγητής ότι έχουμε 50 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή μας. Ναι, 55-50 κάτι τέτοιο λέει ο μιλητή. Ένα προς χίλια δηλαδή, του, το ένα χιλιοστό της, του προπολογισμού της ΚΑΠ. Αυτό για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στον κόσμο θα δώσουμε το ένα της χιλίης. Αυτό είναι σωστό ποσοστό. Αυτό θα φέρει την ανταγωνιστικότητα η οποία μας απασχόλησε δύο ώρες σήμερα ή μήπω θεωρούμε ότι είναι λίγο το ποσό, μικρό το ποσό, μικρό το ποσοστό αυτό. Δεύτερο κεντρικό ερώτημα για αυτό το θέμα. Γιατί, ποιο θα είναι το αντικείμενο της ε, ε, της ε, διαφήμισης, ε, διαφήμισης για κάτι που ήδη υπάρχει στην αγορά. Οι κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση πλέον είναι πάρα πολύ αυστηροί πρέπει να κάνει κανείς ε, ε, πρόθεση για κάτι που υπάρχει ήδη ε, το ευρωπαϊκό μήλο ή το ευρωπαϊκό κρασί ή τα ευρωπαϊκά ζυμαρικά δεν υπάρχουν ακόμα. Υπάρχει το Μπορντό, υπάρχει ο καμπανίτης ίνος της περιοχής Σαμπάνι. Ναι, δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο. Δεν υπάρχει έτσι ένα γενικό προϊόν, ευρωπαϊκό μήλο, ευρωπαϊκό κρασί κτλ. Και επομένως πρέπει να πούμε επίσης ότι οι περισσότερες ε, ε, επιχειρήσεις δεν ξέρουν ακόμα, δεν μπορούν και οι ίδιες να πούν ποιο είναι το, το προϊόν το οποίο θέλουν οι ίδιες να προωθήσουν. Από το αδίέξοδο αυτό μπορούμε να βγούμε εάν βασιστούμε στις ε, ονομασίες προέλευσης, γιατί αυτό αυτές οι ονομασίες προέλευσης είναι ορατές στην αγορά, είναι ευρωπαϊκές ε, ονομασίες ε, ε, ενώ στις, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ιδιωτική ετικέτα θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα. Αυτά είναι τα κυριότερα ζητήματα τα οποία με απασχολούν σε σχέση με αυτή την εργασία. Και βεβαίως μην ξεχνούμε ότι θα έχουμε και ένα νομοθετικό φάκελο τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λουίς Κάπολα Σάντος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα ήθελα απλά και μόνο να ενημερώσω τον εισηγητή και τους συναδέλφους, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψιμες δυσχέρειες για την οικονόμηση, για την ε, χρηματοδότηση αυτών των μέτρων, έλαβα υπόψη το να ενταχθεί αυτή η πτυχή σε σχέση με τις συζητήσεις. Στις προ... επόμενες συζητήσεις θα πούν οι συνάδελφοι αν αυτή η απόφασή μου ήταν σωστή ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λουίς. Ο Διευθυντής, ο κύριος Πατσέκο και μετά ο Ζωζέ Πουδέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή τον Ζωζέ Δεν θα επαναλάβω. Έκανε μία πολύ καλή περίληψη της ανακοίνωσής μας. Πρόθυσε επίσης και μερικές ιδέες οι οποίες τίνουν προς την κατεύθυνση της, του σκεπτικού μας. Πρέπει να προθίσουμε τα συστήματα μας παραγωγής, αηφόρα συστήματα, τις ε, γεωργικές μας πρακτικές, ένα σημείο που ανέφεραν δηλαδή και άλλα μέλη της Επιτροπής και που τίνουν προς την κατεύθυνση που θέλουμε για το πρόγραμμα πρόθεσης. Τώρα, πώς απαντάει κανείς σε μια κρίση. Ε, αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ αργό το σύστημα. Με το σύστημα δηλαδή δήλωση ε, δήλωσης ενδιαφέροντος κλπ. Πώς μπορούμε εμείς σε μια περίπτωση Κρήτης να απαντήσουμε. Πιο γρήγορα και προσθετικά. Τώρα, για τα διάφορα... Για τα κονδύλια. Πού πάνε αυτά τα κονδύλια. Εμείς ε, θα πρέπει στην πρόθεση των προϊόντων να εκρισταθούμε στο ύψος τους. Για τα πιο ειδικά θέματα θέλω να προσθέσω ότι πρέπει να στοχεύσουμε και στην κατάκτηση εξωτερικών αγορών εκτός της Ένωσης και θα πρέπει κατά συνέπεια να φανταστούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μάρκες. Αυτό συμβαίνει για το κρασί. Αλλά θα πρέπει να, φανταστούμε, να το σκεφτούμε και για τη γενικότερη πρόθεση των προϊόντων. Μήπως θα έπρεπε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την εικόνα μας και με μάρκες για να μπορέσουμε να εισχωρήσουμε πιο εύκολα σε τρίτες αγορές. Και ο κύριος Ντόρφμαν προς αυτήν την κατεύθυνση έτεινε. Και έμεσα και η κυρία Πατράου Νέβης. Ο κύριος Εμείς έχουμε ένα 9% του προϋπολογισμού μας που πάει σε προγράμματα αναχώρα. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να μπορούμε να προωθήσουμε ευρωπαϊκά προϊόντα, δράσεις, συστήματα παραγωγής που θα συμπεριλαμβάνουν πολλά προϊόντα και πολλές χώρες. Κύριε Πρόεδρε, μια τελική αναφορά στο γεγονός ότι αναγνωρίζουμε απόλυτα την σημασία του μικρού κυκλώματος. Αλλά αυτό χρηματοδοτείται από τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Θεωρήσαμε, λόγω δηλαδή και των περιορισμένων πόρων, και του τι ρεαλιστικά μπορούμε να προβλέψουμε, θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουμε και με αυτό τον προϋπολογισμό της καμπάνιας πρόθεσης. Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να κρατήσουμε τη χρηματοδότηση μέσω των άλλων προγραμμάτων. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Συμπεράσματα ο Ζωζέ Μποβέ. Άκουσα συνολικά όλες τις σκέψεις, να δούμε πώς θα τις διαρθρώσουμε. Ναι, καταλαβαίνω για τον προϋπολογισμό ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά αν αυτός ο προϋπολογισμός στοχεύει στην πρόθεση των διαφόρων προϊόντων και από την άλλη ανταποκρίνεται και σε περίπτωση κρίσης, ε, τότε θα έχουμε ένα πρόβλημα. Διότι άμα έχουμε και καμιά σημαντική κρίση τότε θα, θα, θα, θα, θα φαγωθεί όλος ο προϋπολογισμός. Άμα θέλουμε εμείς έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό και με μία συνέχεια θα πρέπει να βρούμε πού θα βρούμε τα λεφτά για την κρίση. Θα πρέπει να το σκεφτούμε με την Κομισιόν πώς μπορεί να απαντήσει με έναν ειδικό προϋπολογισμό για τις κρίσεις. Και άμα θα πρέπει να ενσωματώσει στον προϋπολογισμό και την κρίση και να έχει δηλαδή και ένα μόνιμο κονδύλι για την κρίση, δεν θα έχουμε ποτέ προϋπολογισμό. Θα είναι εντελώ κουτσουρεμένος και δεν θα χρησιμοποιηθεί. και δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει να προχωρήσουμε από αυτό. Ένα άλλο σημείο, <coughs> το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να είμαστε σαφέστατοι, όταν μιλάμε πολύ ότι πρέπει να ανοιχθούμε προς τρίτες αγορές, λένε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε μερίδια στην αγορά στις αναδυόμενες χώρες ή σε άλλες. Πρέπει να είμαστε σαφέστατοι. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε εμείς τα διάσημα προϊόντα μας, ε, αλλά όχι να περνάμε τα τρέχοντα προϊόντα τα οποία δεν έχουν εύσημα σε αυτές τις τρίτες αγορές. Δηλαδή θα πρέπει να περνάμε τα προϊόντα τα οποία έχουν ιδιαιτερότητα, όχι εμείς να αντιπαραθέτουμε ε, τα δικά μας προϊόντα με ταυτόσημα τρέχοντα προϊόντα των ε, τρίτων αγορών. Πρέπει να προωθήσουμε τις γεωγραφικές προελεύσεις, τις ανώτατες προελεύσεις κτλ. Διότι εκτός από το κρασί, για όλα τα άλλα προϊόντα, τυριά κλπ, έχουμε περιορισμένα εξαγωγικά μερίδια, ενώ στο κρασί είναι πολύ σημαντική η εξαγωγή του. Αυτές είναι μερικές απαντήσεις για τις τοπικές αγορές και εδώ θα ήθελα να απαντήσω κάτι στην Κομισιόν για να εξηγήσω γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Η ιδέα είναι να πούμε ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι οι τοπικές αγορές οικονομικά και κοινωνικά επιτρέπουν να ε, πουλήσουν οι μικροί παραγωγοί τα προϊόντα τους. Και θα πρέπει λοιπόν να πηγαίνει ο κόσμος να προμηθεύεται τα προϊόντα του στις τοπικές αγορές. Δεν θα πρέπει εμείς να προωθήσουμε όλα τα συστήματα ε, σύντομου κυκλώματος ε, ε ή τοπικών αγορών. Απλώς θα πρέπει να διαρθρώσουμε καλύτερα αυτό το σύστημα ε, τοπικών αγορών που έχει καταστραφεί σε πολλές χώρες όπως είναι η ε, Μεγάλη Βρετανία, οι λαϊκές δηλαδή στην ε, Μεγάλη Βρετανία με φρέσκα προϊόντα που πάνε παραγωγή και τα πουλάνε έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε αυτή την κοινωνική και οικονομική δυναμική. Αυτές είναι μερικές ε, παρατηρήσεις και μετά θα μπούμε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Ζωζέ, ευχαριστώ τους πάντες πέρας της συνεδρίασης. Αύριο το πρωί στις 9 συνεχίζει η Κομαγκρή και στις 3 το θυμίζω συντονιστές και εισηγητές. Θα συναντηθούμε με τον Επίτροπο Τσόλος. Καλό απόγευμα. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εξαιρετικά. Μα, μαγευτικά. Ναι, θα μπορούσα να πω, ναι. Θα Εξωτικά. Να πω. Εξωτικά τα λες, ε. Μαγευτικά. μαγευτικά, μαγευτικά. Παραδείσια. Σαγηνευτικά. Σαγηνευτικά. Όπως έλεγε ο άλλος, είναι πολύ σεξι αυτή η ιδέα. γοητευτικά. Πολύ ωραία. Ε, ναι, κάτι από αυτή την έκθεση που κάνανε αυτή την ε, άλλη, που βρίσκω πολύ σεξι την ιδέα αυτή. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ πάω να κάνω ένα τσιγάρο στο σετνό Ζουαγιές, διότι χαρμένες. Συγγνώμη, ε, στην αργό Ζουαγιές ε, έχει και μια άλλη κονοτάσιο. Α, ναι. Είναι η όχης. Έλα, αλήθεια. Ναι, ναι. Α, δεν το ξέρα. Ε, το ξέρεις, Σιανούλα. Εγώ όχι. Συγγνώμη, όχι. Πολλά γαλλικά ξέρω εσύ. Αυτά τα γαλλικά. Ναι. Αυτά τα γαλλικά. Εμείς που κορίτσια καλών οικογενειών. Εγώ για τις... Εγώ για... ένα ποίημα. Ναι, ναι, το με τις... Ένα πόνημα με πόσες χιλιάδες βέρες. La joyeuse. La joyeuse είναι και ένα κόσμο που έχει να κάνει με τον... Ε, με την είσοδο εδώ των βασιλέων. Όχι στην... Ε, ε, στον πίνακα, σε, σε, αυτόν τον πίνακα του... τον διάσημο πίνακα του Λουί XIV του Ιασίντ ναι. αυτό που κάθεται έτσι. Που κάθεται, ναι, που είναι Α, με το μαλλί. Λοιπόν, λοιπόν, έχεις ε, πάνω στο τραπέζι le Joyeux <laughs> Ε, που δεν είναι τα αρχίδια του βασιλέως. Όχι, συγγνώμη, σου είπα ότι αυτό είναι ε, αργοτίκ, είναι αργό. Ε, ναι, μάλιστα. Δεν είναι... Αυτός... το μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. ναι, εγώ έτσι ναι. έμαθα γαλλικά, κύριε Κάτσε, κατεβαίνεις από ποια πόρτα. Από εδώ έξω. Εγώ θα... Ε, Θα έρθεις να πάρουμε σαν σερ μαζί. Οι τόσες ναι. χιλιάδες βέρς που <laughs> έγραψε αυτός είναι... Κάτι άλλο, δεν είναι βέργες ούτε είναι. είναι ναι, κάτι άλλο. <laughs> Καλό απόγευμα. Παλούκια. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε. Γεια. τι. Επανάληψη ανεπενεργοποιημένη, όχι βέβαια. αξιολογούν. Ναι. Η αφύπνιση αποθηκεύθηκε Μάλιστα. Όχι ρε, γαμώτο, στο διάλογο πια.